Έχουμε την τροπολογία υπαριθμό 3. Είμαστε στην έκθεση της κυρίας Κέλλερ. Η τροπολογία 3 της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έτσι δεν είναι. Amendment number 10, made also by... Η 10, πάλι τη σύνταξη, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 12, υπέρ. Πάντα τη σύντα, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η προφορική τροπολογία υπαριθμών 1 της κυρίας Κέλλερ. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η προφορική η δύο, πάλι Κέλλερ. Α, εμείς διαφωνούμε με την προφορική αυτή τροπολογία, αλλά δεν μπορούμε να τη θέσουμε σε ψηφοφορία. Η παριθμό 3 τότε, πάντα προφορική, το ίδιο. Το αυτό, καλά, δεν την ψηφίσουμε τότε. Η 26 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 27. Έχει ζητηθεί από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ε, ψηφοφορία κατά τμήματα. Τμήμα πρώτο, υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 28 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 ψήφι υπέρ κατά αποχές Φαίνεται σαν να έχει απορριφθεί, αλλά δεν ξέρω πάλι. 30. Who is in favor? 30 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 9 ίντα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 11. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική υπαριθμών 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές μάλλον θα χρειαστεί κάποιος έλεγχος, ενδεχομένως. Η ηλεκτρονική απολύθευση Αλλιώς είπε τα χέρια να σας ξαναμετρήσουμε. Τη συμβαστική υπαριθμό, ναι. Κατά. So 12 to 9, εγκρίνεται. We άλλο έλεγχο θέλετε. Who is in Και τρίτος έλεγχος. Υπέρ. 12... υπέρ, είπαμε και πριν 12 είσαστε. 13 τώρα. Με μένα. against? Κατά. 13 10 adopted. 13-10 εγκρίνεται. Η 31 καταπίπτει μάλλον. Η 32 έχει αποσυρθεί. Η συμβαστική μόνο 2. Ψήφι πέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 κατά πίπτη μάλλον έτσι. Μάλιστα. Ή 34 ψήφι πέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ή 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η προφορική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 36 καταπίπτει. 37 υπέρ. Κατά. Έλεγχος χρειάζεται και πάλι εδώ. Ψήφι πέρα. Δεκατρεις. Κατά. Έντεκα. Εγκρίνεται λοιπόν. Η 38 ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. Η προφορική υπαριθμό 5. Ψήφι Κατά. Με την ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. Η 39 καταπίπτει. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 41 έχει αποσυρθεί. Η προφορική υπαριθμό 6 ψήφι πέρα. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Η 42 της κυρίας Τόια. Ψήφι πέρα. Κατά. Δεκατέσσερα δώδεκα εγκρίνεται. Η προφορική υπαριθμό 7. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 κατά πίπτη. Και συνεχίζουμε. Συμβαστική ή υπαριθμό 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 κατά πίπτη 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, η προφορική υπαριθμών 8 ψήφι υπέρ. Όχι, δεν ψηφίζουμε 9. Ε, ούτε. 46 ε, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 47 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική αριθμών 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Α, όχι, όχι, έχει καταπέσει. Και η 49. Όλες μέχρι και την 51. Και πάμε στην και 52 έχει προσθεθεί 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβιβαστική υπαριθμών 5. Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Αχ, έχει καταπέσει. Πάμε στην 58 κατευθείαν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 59 καταπίπτει. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε μία γλωσσική που δεν την ψηφίζουμε. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική υπαριθμό 6. Η υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 καταπίπτει. 63 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η προφορική υπαριθμό 10 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64. Καταπίπτει. Η παράγραφος 10 ε, ξεχωριστά ψηφίζεται υπέρ, κατά, οι σοσιαλιστές το έχουν ζητήσει αυτό, να ψηφιστεί χωριστά από αποχές. Απορρίπτεται, έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Η προφορική τροπολογία τώρα υπαριθμών 11. Υπέρ. Έχετε αντίρρηση. Έχετε εντύπωση ή δεν έχετε, αποφασίστε. We don't take it. Άρα δεν την ψηφίζουμε. Καλώς. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68 υπέρ. Υπέρ. 68 παρακαλώ. Κανείς δεν είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 69, 70 και 71 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά εγκρίνεται η προφορική τροπολογία υπάρχει 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει. Η συμβαστική 7 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 74 καταπίπτει. Έχουμε χωριστή ψηφοφορία που ζήτησαν οι πράσινοι. Κατά τμήματα μάλλον. Και ίντα 1 υπέρ του πρώτου τμήματος της ίντα 1 κατά αποχές έλεγχος Squeeze in favor. Υπέρ, τα χέρια σας. Κατά. Μάλλον εγκρίνεται. Φαίνεται. Το δεύτερο τμήμα είναι τα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μάλλον έτσι δεν είναι το πρώτο τμήμα της 2 υπέρ πάντα τη σύντα κατά αποχές εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Εγκρίνεται. Η προφορική υπαριθμών 13. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Το επόμενο καταπίπτει. 8 της είναι τα ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 75 έχει αποσυρθεί. Η 76 είπε Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 77 κατά πίπτη. Η 19 ίντα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 78 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 81 έχει, απορριφθεί, έχει αποσυρθεί, συγγνώμη, 82 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Είναι τα 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα υπαρθών 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται είναι τα 22 ψηφιπέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ίντα υπάρχουν 13. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ίντα 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ίντα 15. Υπέρ. Κατά. Πώς είπατε. Κατά παρακαλώ. Αποχές εγκρίνεται. 85 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 90. Καταπίπτει. 91. Καταπίπτει. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93. Καταπίπτει. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Είναι τα 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα 18. Ορίστε. Α, υπάρχει μια πρόταση εδώ να ψηφιστούν μαζί οι 18 μέχρι και την 24. Ψηφιπέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παίρνουμε αμέσως στην 96 ψήφι Κατά. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 8 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον απορρίπτεται έτσι φαίνεται. Θέλετε να ξαναψηφίσουμε υπέρ της συμβαστικής παρελθόν 8 παρακαλώ. κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική εννέα ψήφι Κατά. αποχές εγκρίνεται. 100, όχι, επόμενες καταπίπτουν. Directly to 100. Πάμε ε, κατευθείαν στην 103, ψήφι πέ. Κατά, αποχές, μάλλον εγκρίνεται. 104, ψήφι πέ. Κατά, αποχές έχει απορριφθεί. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10 είπε. Κατά. Εγκρίνεται. 105 καταπίπτει. 106 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η προφορική 14 ψήφι υπέρ. Υπέρ της προφορικής 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν κρίνεται έτσι δεν είναι. Τότε να πάμε στην 112. Ψήφι Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά δεν είμαι σίγουρη. 112 είπε. Κατά. Δώδεκα έντεκα είναι δεν είναι 12-12. Να ξαναψηφίσουμε. Κατά. Τα κατά. Δώδεκα δεκατρία απορρίπτεται. 117. Όχι, 113, συγγνώμη. 113, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 Είπε κατά εγκρίνεται 115 Είπε κατά αποχές εγκρίνεται 116 Είπε κατά αποχές απορρίπτεται 117 είπε κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 11 καταπίπτει και πάμε στη 13 του κυρίου Γκέρνς, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ υπέρ είπα κατά απορρίπτεται 18 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 19 υπέ, κατά εγκρίνεται 20 υπέ, κατά εποχές, εγκρίνεται η προφορική 15 δεν διαφωνεί κανείς να ψηφιστεί ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίφτεται 22 υπέρ. ΑΤΑ, Αποχές. γκρίνεται. Δηλαδή, έλεγχος. <laughs> Ψήφι υπέρ της 22 ή 22. Κατά. Abstentions. Adopted. Αποχές εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πού είμαστε τώρα. 24. 24 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πέντε υπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα τι έχουμε. Ψηφίσουμε όλες μαζί, όλες μέχρι το τέλος. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται το σύνολο. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να ψηφίσουμε την ε, γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές. Εγκρίθηκε και η γνωμοδότηση στο σύνολό της και σας ευχαριστώ. So congratulations to the rapporteur. Συγχαρητήρια στην κυρία Κέλλερ, την εισηγήτρια. Πάμε καλά. Πάμε στις αγορές των παραγόγων. Πάμε στη δεύτερη σημερινή έκθεση, μελλοντικές ε, δράσεις πολιτικής με συντάκτια την Εύα Ζολή. Τέταρτη τροπολογία υπέρ. Περάσαμε στην επόμενη έκθεση. Ποιος είναι υπέρ της ανατροπολογίας 4. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 5. Τροπολογία 5. Το ΕΛΚ ζήτησε χωριστή ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογή υπαριθμών 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Έχουμε την 7 μαζί με την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Ψηφίζουμε την 1 και τη 2 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τρίτη τροπολογία. Μαζί με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και τώρα ψηφίζουμε συνολικά την γνωμοδότηση υπέρ, κατά, αποχές. Υιοθετείτε. Συγχαρητήρια κυρία Ζολή So, we move now on. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο. So we can continue. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Uh, colleagues, uh, we can move on democratic scrutiny of programming. Πάμε στο δημοκρατικό έλεγχο του προγραμματισμού στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την ανάπτυξη. Παρουσίαση των περασμάτων των ομάδων εργασίας, ε, ανταλλαγή απόψεων και ενδεχομένως συστάσεις. Τις τελευταίες εβδομάδες Λάβαμε από την Κομισιόν μια σειρά από έγγραφα στρατηγικής ε, για την εφαρμογή του DCI ε, που εξέτασαν οι διάφορες ομάδες εργασίας. Ο Noise Searcher από την ομάδα εργασίας Α ε, δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα. Γι' αυτό εγώ πρέπει να παρουσιάσω τα αποτελέσματα για τη Μογγολία, τις Φιλιππίνες. I will make a short briefing uh, on behalf of Mr. Θα κάνω μία μικρή παρουσίαση για τη Μογγολία ομάδα εργασία Α, ε, αξιολόγηση του, της ενδιάμεσης έκθεσης για το έγγραφο στρατηγικής ε, της ε, χώρας αυτής. Οι συζητήσεις έγιναν για την κατανομή 8 εκατομμυρίων στις μογγολικές αρχές για να δημιουργήσουν το δυναμικό για να ευθυγραμμιστούν με τα πρότυπα DCI της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν δράσεις σε διάφορους τομείς στο πλαίσιο της, του εμπορίου, της περιφερειακής ολοκλήρωσης, ε, επενδυτικά μέτρα για το εμπόριο, τεχνική βοήθεια και δημιουργία δυναμικού για να εφαρμόσουν και να προωθήσουν ε, υγιείς πολιτικές. Ε, υπάρχουν πολιτικές που δεν συνάδουν απόλυτα με το DCI ε, και με τους τομείς DAC. Γι' αυτό λοιπόν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να γίνουν κάποιες αλλαγές ούτως ώστε να γίνουν σεβαστό ε, και οι τομείς DCI ε, και οι τομείς DAC. Παραδείγματο χάρη βοήθεια για να εφαρμοστούν υγιείς εμπορικές πολιτικές. Θα πρέπει το αναθεωρημένο κείμενο να αναθεωρηθεί προς την κατεύθυνση της εφαρμογής αυτών των προτύπων από τις μογγολικές αρχές. Και πρέπει να, για τις δραστηριότητες δύο θα πρέπει να γίνει σεβαστό το DCI, προκειμένου η Μογγολία να ενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία. Η ομάδα εργασίας Α προτείνει με βάση το άρθρο 37 του DCI να περάσει το έγγραφο αυτό από τη διαδικασία της επιτροπολογίας. Θα μιλήσω για τις Φιλιππίνες. Η ομάδα εργασίας Α ε, εκτιμά ότι η ενδιάμεση έκθεση για το έγγραφο στρατηγικής των Φιλιππινών απαντάει σε διάφορα μελήματα και ανησυχίες ε, του εισηγητή ε, για τις δραστηριότητες ε, που, του κατά πόσον δραστηριότητες μάλλον αυτές συνάδουν με τον κανονισμό DCI. Ε, η ομάδα της Μογγολίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζήτησαν διάφορα θέματα γιατί παραδείγματο χάρη έχουν παραμελήσει τον τομέα της εκπαίδευσης και γιατί κάποια κονδύλια από την εκπαίδευση πηγαίνουν στην υγεία. Θέλουμε και εμείς να συμμετάσχουμε ενεργά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις συζητήσεις ε, και στις συζητήσεις με τους stakeholders για τη σύνταξη του, της ενδιάμεσης έκθεσης. Ε, υπάρχει ανισορροπία στη χρηματοδότηση, ε, στην, ε, στις βασικές υπηρεσίες και στις υγείες ε, και γενικά ε, παραμελείται ο τομέας της εκπαίδευσης. Ε, όμως ε, η δικαιολογία των αρχών είναι ότι ο τομέας της ε, εκπαίδευσης καλύπτεται από τα κονδύλια άλλων δωρητών. Δεύτερον, ε, για τις ενευτικές συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε οποιαδήποτε εξέλιξη να μας βρει σύμφωνος, δηλαδή θα πρέπει να εμπλακούμε. Η Ισπανία και η Γερμανία και ο ILO και η UNICEF ε, συναντήθηκαν και συζήτησαν με τις αρχές των Φιλιππίνων ε, στα πλαίσια των διαβουλεύσεων αυτών. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση από την Κομισιόν σε θέματα διαφθοράς, λέει η ομάδα εργασίας. Η ομάδα εργασίας Α λέει ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία Η ομάδα εργασίας Α δεν είναι αντίθετη με το έγγραφο ε, για τις Φιλιππίνες ε, με βάση τα όσα προβλέπει το άρθρο 35 ε, του DCI. Συνάδελφοι, συμφωνείτε με τις συστάσεις της ομάδας εργασίας Α για τη Μογγολία και τις Φιλιππίνες. Αν ναι, Θεωρώ ότι η Επιτροπή έχει υιοθετήσει τις συστάσεις. Υπάρχει και προθεσμία, ε, ή μάλλον έχει ολοκληρωθεί η προθεσμία για το δικαίωμα ελέγχου. Τώρα για το Λάος. Η κυρία Θεοχάρους για το Λάος. Thank you very much. Thank you, Madam Chair. Η ομάδα εργασία Α αξιολόγησε την ενδιάμεση αναθεώρηση στη συνεδρίαση που έγινε την 31η Μαρτίου θεωρήσαμε ότι η αξιολόγηση για τη συνεργασία του 2008 είναι θετική γιατί τονίζεται ότι ε, στήριξε δημοσιονομικά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες ε, και ε, εκφράσαμε την υποστήριξη μας για τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική στήριξη με σαφή σαφέστατε συνθήκε σχετικά με τη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση που θα δοθεί στο λαός μόνο αν καταδειχθεί η πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της υγείας και τη εκπαίδευση. Λυπούμεθα που ε, το πρόγραμμα για τη διατήρηση και για την ασφάλεια, η εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών παρουσιάζουν, ε, ε, ε, εξακολουθούν να παρουσιάζουν προβλήματα στο λαός. Δεν υπάρχουν μέτρα και διαδικασίες που θα εξασφαλίσουν ας πούμε, την υλοποίηση πολιτικών για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας. Υπήρξαν σημαντικές πρόοδοι για την καταπολέμηση για την παροπλισμό μάλλον βομβών που δεν έχουν ακόμη εκραγεί. Βέβαια, θα θέλαμε περισσότερε πληροφορίε σχετικά με το ποσοστό του εδάφους που πλήττεται και ε, ποιο ποσοστό του εδάφους έχει ήδη, ε, είναι ελεύθερο και έχει καθαριστεί από αυτέ τι βόμβες. Ε, θεωρούμε ότι προς το παρόν οι απαντήσεις ε, δεν επαρκούν, αλλά δεν αντιτασσόμεθα στην ενδιάμεση αναθεώρηση ε, βάσει της διαδικασίας επιτροπολογίας που προβλέπεται από το άρθρο 35 της Διαθεσμικής Συμφωνίας. Συμφωνείτε με τις συστάσεις της κυρίας Θεοχάρους. Εγκρίνονται έτσι οι συστάσεις από την Επιτροπή και για το δικαίωμα ελέγχου ε, ε, ε, ορίζουμε την καταληκτική ημερομηνία. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κάσμερα για την ομάδα εργασίας ε και τον κύριο Κασόλη για την ομάδα εργασίας γ. Ο κύριος Κάσμαρ. Η ομάδα εργασίας Β ε, ενδιάμεσα ε, συζήτησε για τον Μπαγκλατές, ε, τη Σρι Λάνκα, το Μπαγκλαντέ, πρώτα η ομάδα εργασίας ΕΒΙΤΑ ικανοποιήθηκε από την ενδιάμεση έκθεση παρά τι ατέλειες ε, που ε, ανακοινώνονται για το 2007, δηλαδή ε, οι ατέλειε που είχαν εντοπιστεί για την περίοδο 2007-2014 έχουν καλυφθεί και επίσης σημειώνουμε καλή στόχευση ω προς τους Δικαιούχου των προγραμμάτων ακόμη και για τι πιο ευάλωτες πληθυσμιακέ ομάδες αυξάνεται, αυξάνεται όμως η διακύμανση των τιμών στα τρόφιμα, τα καύσιμα και στο, ε, οι γραμμές του DCI καλύπτονται και εμπλέκονται περισσότερο οι εταίροι, οι κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία των πολιτών, το Εθνικό Κοινοβούλιο στο Μπαγκλαντές. Η ενδιάμεση αναθεώρηση έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και τη διαχείριση των δημοσίων πόρων, ε, όμως δεν υπάρχουν επαρκή κονδύλια για την επιστημιστική ασφάλεια, η οποία όλα και περισσότερο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στα, ε, σε όλα τα προγράμματα σχετικά με την εξωτερική βοήθεια. Η έλλειψη τροφίμων ε, δεν έχει καλυφθεί επαρκώς. Επίσης, ε, ε, ως δεν επικουρούνται επαρκώς οι πρόσφυγες στη βάση της αρμόδιας πολιτικής για τις κλιματικές αλλαγές. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ειδικά στοχευμένα μέτρα για την ανάπτυξη και την βοήθεια. Η στρατηγική μας μέχρι τούδε επικεντρωνόταν στον εξαγωγικό τομέα, αλλά δεδομένου του στόχου της μείωσης της στόχια, και το πιθανό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στους βασικούς εξαγωγικούς τομείς, θα έπρεπε να στηρίξουμε όλους τους εξαγωγικούς τομείς. Συστήνουμε στην Επιτροπή ΝΤΕΒΕ να μην ενταχθεί στο CSP, στην ενδιάμεση αναθεώρηση δηλαδή για το Μπαγκλαντές. Αυτό είναι το τελικό μας ε, πόρισμα, είναι θετικό. Τώρα, ε, ε, εκτιμούμε το ότι ε, η στρατηγική εστιάζεται πλέον στο θέμα της διακυβέρνησης, ούτως ώστε η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διοχετευτεί στο περιβάλλον, στην καταπολέμηση του λαθρομπορίου ναρκωτικών και στην ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης, δεδομένη της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τις κλιματικές αλλαγές. Είναι ικανοποιητικά, ικανοποιητικές οι προτάσεις, αλλά δεν υπάρχουν επαρκή κονδύλια για ε, μόνο 6 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2011-2014. Σε βασικούς τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση δεν είναι ικανοποιητικά τα αποτελέσματα επειδή υπάρχουν λιγοστά κονδύλια. Μας ανησυχεί επίσης το ότι δεν αναφερόμαστε στις διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών ή με την Εθνική Βουλή ε, ε, για την περιφερειακή συνεργασία ε, θεωρούμε ότι ήταν καλά τα αποτελέσματα και έχει ενσωματωθεί και η μήτρα των στόχων της χιλιετίας, ε, το οποίο βρίσκουμε ικανοποιητικό. Η ομάδα εργασίας Β προτείνει προς την ε, Επιτροπή Ανάπτυξης να μην αντιταχθεί στην διάμεση αναθεώρηση με τις ε, Μαλδίβες. Τώρα, ε, κατόπιν υπήρξε επικαιροποίηση των δεδομένων ε, για την κατάσταση που επικρατεί επί τόπου και ε, πρέπει να διατηρήσουμε την προσέγγιση που βασίζεται σε πιθανά σενάρια. Δύο είναι τα πιθανά σενάρια που θα προσαρμόζονται κατά τη διαδικασία αναθεώρησης. Σε πρώτο σενάριο, συμφιλίωση στην Σρι Λάγκα ε, σενάριο 2 συνεχίζεται η ανθρωπιστική κρίση και οι συγκρούσεις. 60 εκατομμύρια ευρώ ε, προβλέπονται ε, για την ε, περίοδο 2011-2014 και τα 54 από αυτά θα διοχετευτούν στην ανοικοδόμηση. Κατά τα λοιπά θα χρησιμοποιηθούν για το εμπόριο και για την καλή διακυβέρνηση. Τα περισσότερα προτινόμενα προγράμματα εστιάζονται στο στόχο της μείωσης της φτώχειας. Βέβαια, στο δεύτερο, το, η επιλογή του σενάριου θα επηρεάσει και τη φύση των προγραμμάτων. Αν υπάρξει πολιτική συμφιλίωση, οι δραστηριότητε θα ακολουθούν μια σαφή εντολή. Όμω, ε, βάσει του σενάριου 2 θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες των πλέον ε, ευάλωτων πληθυσμιακών ε, ομάδων. Οι βασικοί τομεί θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την ανάπτυξη της ικανότητας ΕΝΤΑΚ και άρα προτείνουμε στην Επιτροπή να μην αντιταχθεί στην ενδιάμεση αναθεώρηση για τη Στριλάνκα. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να συμφωνήσετε αγαπητοί συνάδελφοι με τις συστάσεις ε, του κυρίου Κάσμαν. Ε, ωραία, έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή οι συστάσεις και έχει περάσει η προθεσμία ε, για το δικαίωμα ελέγχου. Τώρα το λόγο έχει ο κύριο Σασόλη για να μας ε, αναφέρει τα πορίσματα της ομάδας εργασίας ΓΑΜΑ. Με μικρόφωνο κατά προτίμηση. E το θέμα του ownership της ιδιοκτησίας είναι πολύ σημαντικό ε, για να είναι αποτελεσματική η βοήθεια και να υπάρξει πολιτικός διάλογος μεταξύ των δύο μερών. Η κατάσταση ε, έχει διαφυλαχθεί αλλά και βελτιωθεί με το έγγραφο της Εθνικής Στρατηγικής. Η ομάδα εργασία ΓΑΜΑ ε, εκτιμά το ενδιαφέρον που έδειξε η Κούβα για την επανεργοποίηση των σχέσεων και ο πρέσβης της Κούβας έδειξε ότι είναι ικανοποιημένος για το γεγονός ότι το έγγραφο στρατηγικής εθνικής στρατηγικής ε, ασχολήθηκε με τομείς ε, όπως ε, περιβάλλον, επιστηστική ασφάλεια, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ανταλλαγές, κατάρτιση, εκπαίδευση ε, με βάση τις προτεραιότητες που έχουν και οι ίδιες οι κουβανικές αρχές. Ε, κατά την άποψή μας, τα όσα έχουν γίνει από το 2008 και μετά θα πρέπει να οδηγήσουν στην εξομάλυνση των σχέσεων με μια διμερή συμφωνία ανάλογη με αυτή που έχει υπογραφτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, με άλλες χώρες της περιοχής. Η συνεργασία με τη χώρα θα πρέπει να προχωρήσει παράλληλα και αυτόνομα από τις πολιτικές συνομιλίες διμερούς χαρακτήρα που ε, είναι να εξελίξει σήμερα. Κατά την άποψή μα, οι τράσει για την επιστημιστική ασφάλεια, η προσαρμογή στι κλιματικέ αλλαγέ και η βελτίωση των αρμοδιοτήτων ε, για την ανάπτυξη συνάδουν με τους βασικούς μας στόχους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ε, μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας. Η ομάδα εργασίας επίσης εκτιμά την προτεραιότητα που δίνεται για την βιωσιμότητα του κλίματος, αλλά θεωρεί ότι περαιτέρω μέτρα για να μειωθούν οι επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με επιπλέον κονδύλια πολύ πάνω από τους πόρους που έχουν προβλεφτεί και έχουν ε, τεθεί στο, στην άκρη μέχρι στιγμής για την εξάλληψη τη ε, φτώχεια και ο στόχο θα πρέπει να είναι η υλοποίηση των στόχων τη χιλιετίας. Επίσης, ε, εκφράζουμε την ανησυχία μας για την επιδείνωση των δικτών υγείας και θέλουμε η Κομισιόν να ασχοληθεί στο μέλλον με αυτόν. Ε, από το 1996 διάφορες αρρώστιες όπως το AIDS έχουν αυξηθεί αυτό το διάστημα, δηλαδή μέσα σε 15 περίπου χρόνια, ιδίως μεταξύ των ομοφιλοφίλων. Θα πρέπει να ε, καταπολεμήσουμε το AIDS ε, και όμως οποιασδήποτε διακρίσεις, και διακρίσεις ε, ε, υφίστανται αυτές οι ομάδες των ομοφιλοφίλων για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας. Έχουμε τέσσερα βασικά συμπεράσματα. Μετά από πέντε χρόνια αδιέξοδου στις σχέσεις Κούβας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το στρατηγικό έγγραφο προβλέπει μία απορία για τις αμοιβέ μας σχέσεις που θα πρέπει να ενδυναμωθούν. Τα μέλη της ομάδας εργασίας. Ακριβώς γι' αυτό εκτιμούν τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Κούβας και θα πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα και ανεξάρτητα από τον πολιτικό διάλογο που η χώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν σε υπουργικό επίπεδο. Δεύτερο σημείο. Εκτιμούμε την ε, πρωτοβουλία της Κομισιόν να, δουλέψουμε σε τομείς κλειδιάς που έχει καθορίσει η χώρα αυτή. Ε, εκτιμούμε ότι το εστιακό σημείο που είναι η, δυνατότητα των, ε, η βελτίωση της δυνατότητα για ανάπτυξη θα πρέπει να εστιαστεί στην κατάρτιση σε επισκέψεις των εμπειρογνωμόνων για να ενημερωθούν για θέματα ανάπτυξης ε, και να αυξηθεί το δυναμικό της Κούβας για την ανάπτυξη. Θα πρέπει να υπάρξουν και νέες πρωτοβουλίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως ε, και για τα δικαιώματα των ε, γυναικών, ε, δικαιώματα πολιτιστικά, δικαιώματα των ανηλίκων και δικαιώματα σεξουαλικών επιλογών. Το Ευρωπαϊκό Εργαλείο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα υπάρχει στη διάθεσή μας για να υποστηρίξει πρωτοβουλίες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέταρτο σημείο, Παρά τις προσπάθειες αυτές που έχουν γίνει, η ομάδα εργασίας ΓΑΜΑ ζητάει ο ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και την κοινή ασφάλεια να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις σημερινές δραστηριότητες στον τομέα αυτό. Ιδίως μετά τα τελευταία ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κούβα να μα ενημερώσει επίση και για τι μελλοντικέ δράσει που πρόκειται να εφαρμοστούν. Σε αυτή τη φάση τη διαδικασία η ομάδα εργασία συστήνει η Επιτροπή για την Ανάπτυξη να μην θέσει αντιρρήσει για αυτό το εθνικό στρατηγικό κείμενο. Ευχαριστώ και εγώ σα ευχαριστώ κύριε Σασόλη. Ε, ε, συμφωνούμε λοιπόν με τις συστάσεις ε, που μας παρουσίασε ο κύριο Σασόλη από την ομάδα εργασίας Γ. Θεωρώ ότι αυτές οι συστάσεις έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή και έχει κλείσει και προθεσμία για το δικαίωμα ελέγχου. Και τώρα περνάμε στο σημείο 14, στον τριμερή διάλογο για το σχέδιο προεπολογισμού 2011, ο κύριος Θέσμπερμαν είναι ο εισηγητής για το 2011. Είναι η πρώτη διαδικασία κατά του προπολογισμού δυνάμει των νέων κανόνων τη συνθήκη Λισαβόνα. Ε, θα εγκρίνει ψήφισμα για το σχέδιο προπολογισμού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, είναι σημαντικό το ψήφισμα του Κοινοβουλίου διότι θα θέσει τις προτεραιότητες ε, και ε, θα ορίσει την εντολή για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβουλίο στον τριμερή διάλογο που θα γίνει τον Ιούνιο. Είναι σημαντικό να ακουστεί η φωνή της Επιτροπής μας στην όλη διαδικασία. Ο κύριος Μπέργμαν, ο εισηγητής μας, έχει προετοιμάσει μια γνωμοδότηση, την έχετε πάρει στα αγγλικά και στα γαλλικά. Δυστυχώς ε, δεν είχαμε χρόνο για να μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες, αλλά το ταχύτητα το δυνατόν θα σας τη στείλουμε με email. 12 ε, Μαΐου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες, δεν έχουμε πολύ χρόνο δηλαδή στη διάθεσή μας ε, και μέχρι τις 3 Μαΐου θα έχουμε χρόνο για την υποβολή τροπολογιών και μετά θα ψηφίσουμε στις 10 Μαΐου. Ο κύριος Τάις Μπέρκμαν, ο εισηγητής, ε, θα μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπατε σωστά, σήμερα βέβαια το σχέδιο ε, προπολογισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι τον Ιούνιο θα συζητήσουμε το Συμβούλιο και έχουμε και ε, προγραμματίσει ψήφισμα ε, για την Ολομέλεια. Θα πρέπει να δώσουμε το στίγμα μας εκεί για την αναπτυξιακή βοήθεια παρά την κλιματική αλλαγή, τους στόχους χιλιετίας και την οικονομική κρίση Πιστεύω στεναρά ότι έχουμε να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Α ελπίσουμε ότι μπορούμε να πείσουμε και του συναδέλφου του προπολογισμού να ακούσουν τι προτάσει μα καλύτερα από την περασμένη φορά όταν αποφάσισαν να μην υιοθετήσουν καμία από τι δικέ μα συστάσει. Αυτό ήταν το ένα για τη γνωμοδότηση τώρα πάμε. Κλιματική αλλαγή. Έχει προκληθεί από τις βιομηχανισμένες χώρες και πληρώνουν την ύφη φτωχές χώρες. Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα έχουν 100 δις ε, ε, ευρώ το χρόνο σύντομα να πληρώσουν ως λογαριασμό. 2,4 ε, για τη... το μετριασμό και τη μείωση της κλιματικής αλλαγής είναι σημαντικό μεν, από το τίποτα καλύτερο φυσικά για τα μικροδάνεια, για την επιστηστική ασφάλεια. Η κρίση του 2008 όθησε πολλούς ε, ε, στη φτώχεια και στην πείνα. Και έχουν, έχουν ε, ξεπεράσει πλέον το 1 δισεκατομμύριο εκείνοι που υποφέρουν από την πείνα. Καλά είναι τα μικροδάνεια και οι μικροπιστώσεις για να βοηθούν μικρούς παραγωγούς, κυρίως γυναίκες, για να είναι αυτάρκοι σε τρόφιμα και να έχουν επιστηστική ασφάλεια. Το 2009-2010 είχαμε προϋπολογισμούς που υποστήριξαν τέτοια σχήματα και τονίζουμε την ανάγκη να συνεχιστούν αυτά και να επεκταθούν. Επίσης, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τον προϋπολογισμό για να δώσει καλύτερη προτεραιότητα σε πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στι αναπτυσσόμενες χώρες, πρόσβαση σε δάνεια, σε αποταμιεύσεις, σε συστήματα ασφαλίσεων ε, ε, για την υγεία των προσώπων αλλά και να ασφαλίζουν και τις οδιές του. Το εργαλείο τώρα αναπτυξιακής συνεργασίας, DCI, με ε, βρίσκει αντίθετο απολύτω, όπως και πολλούς συναδέλφους, να παίρνουν κονδύλια από εκεί για να τα πηγαίνουν αλλού. Οποιαδήποτε μεταφερά πιστός, οποιαδήποτε νομική βάση και αν επικαλεστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έρχομαι στην πρόταση ICI Plus και ε, κυρίω για τις χώρες ΑΚΕ που παράγουν μπανάνες. Δεν ξέρω αν χρειάζεται υπενθύμηση. Θυμίζω πάντως ότι το ε, μέσο αυτό ε, έχει στόχο να μειώσει τη φτώχεια και όχι να ενισχύσει τις καλές μας σχέσεις με ε, χώρες ευημερούσες. Το Συμβούλιο έρχεται με μια νέα πρόταση και πάλι μια καινούργια πρόταση ακολουθεί την προηγούμενη. Έχει πολλές φιλοδοξίες, αλλά λεφτά δεν έχουμε για τις φιλοδοξίες του Συμβουλίου η αναπτυξιακή ε, πολιτική δεν θα πρέπει να πληρώσει την ύφη αυτής της όρευσης νέων ε, πρωτοβουλειών. Αφήστε δε που είναι και λίγο το προσωπικό, ε, πολύ λιγότερο από τους άλλους διεθνείς δωρητές για την αναπτυξιακή βοήθεια. Εγώ δεν θέλω να υπερασπιστώ καμία γραφειοκρατική μηχανή, αλλά θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε προσωπικό ε, που να εκτελεί σωστά επιτόπου ε, τις πολιτικές που εμείς αποφασίζουμε. Δηλαδή να έχουμε και τα μέσα τα οικονομικά που να μας επιτρέπουν να ε, εκτελούμε σωστά αυτές τις πολιτικές. Επαναλαμβάνω, ζητώ και πάλι απλούστευση των διαδικασιών για ε, βοήθεια βιώσιμη, προβλέψιμη και καινοτόμε ε, μορφές και πηγές χρηματοδότησης τη αναπτυξιακή βοήθειας. Αυτός είναι ο κύριο κορμός λοιπόν της νομοδότησή μου. Ε, περιμένω ανυπόμονα να ακούσω και τις δικές σας προτάσεις και το σχέδιο προπολογισμού μόλι σήμερα εκδόθηκε κυκλοφόρησε. Αφού μελετήσω τα στοιχεία θα έρθω και σε τεχνικές μάλλον λεπτομέρειες για να προσαρμόσω και το κείμενο στην πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τα ενδιαφέροντα και ξεκάθαρα σχόλιά του κατά την εισαγωγική του παρουσίαση. Όπως είπε, το σχέδιο προϋπολογισμού δημοσιεύθηκε σήμερα και μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού δημοσιεύουμε και μία έκθεση για την λειτουργία της Διαθεσμικής Συμφωνίας. Ε, μας τα λόγια όταν το λέω. Η έκθεση, γενικώς πώς, αναγνωρίζει την χρησιμότητα της σημερινής ε, δημοσιονομικής διαδικασίας. Το σημερινό πλαίσιο πολιετές ε, για τη χρηματοδότηση λειτουργεί από ό,τι φαίνεται αρκετά καλά. Είναι αλήθεια ότι ο τίτλος 4 πάντα είναι υποπίεση. Το ξέρουμε, γιατί μας ζητάνε συνέχεια να ανταποκριθούμε όχι μόνο σε καταστροφές και θεομηνίες, και αυτό δημιουργεί προκλήσεις και προβλήματα σε άλλους τομείς, αλλά γενικώ ε, πώς καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε πολλές καταστάσεις. Ε, αυτό είναι το πλαίσιο, όπως λέει και ο εισηγητής, ε, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούμεθα και κινούμεθα. Ανέφερε επίσης τα συνοπτικά μέτρα για την μπανάνα. Εκεί χρειάστηκε να εξετάσουμε διάφορες δυνατότητες για χρήση μέσων από άλλους τομείς στα πλαίσια της διαθεσμικής ε, συμφωνίας. Ούτως ώστε τα χρηματοδοτικά μέτρα, τα συνοδευτικά μάλλον μέτρα για την μπανάνα να προωθηθούν ε, χάρη στην ευελιξία. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες για το DCI, το μέσο για την αναπτυξιακή συνεργασία, αλλά μην νομίζετε ότι μειώνουμε τα ανώτατα όρια ε, τα οποία είχαμε συμφωνήσει. Αντίθετα, ε, στην περίοδο 2007-2013 έχουμε προσθέσει 400 εκατομμύρια ευρώ. Δεν παίρνουμε χρήματα, αντίθετα, βάζουμε. Αν συγκρίνεται το πρώτο χρόνο του 2000, ε, της περίοδου 2007 ε, με το 2013 υπάρχει μια αύξηση κατά 26%. Σημαντική αύξηση στα κονδύλια, έτσι. Ε, τώρα πάμε στις μικροπιστώσεις και στην επιστημιστική ασφάλεια. Οι σημερινές δραστηριότητες ε, υπό την ε, γραμμή του προπολογισμού την πιλωτική ήταν πολύ χρήσιμη. Το 2009 χρηματοδοτήσαμε ένα πρόγραμμα στην Παλαιστίνη και στην Αϊτή. Παρότι το πρόγραμμα στην Αϊτή βεβαίως ε, καθυστέρησε λόγω των προφανών προβλημάτων που είχαμε και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δεσμεύσουμε τα κονδύλια του 2010. Ε, για τη διευκόλυνση για τα τρόφιμα υπήρχαν νέα, προγράμματα για μικροπιστώσεις που εγκρίθηκαν ε, για τη διευκόλυνση των τροφίμων και στο μέλλον ε, συμπεριλαμβάνουμε και τις μικροπιστώσεις στα πλαίσια της πολιτικής για την επισητιστική ασφάλεια. Επομένως δεν υπάρχει ανάγκη για μια πιλωτική δημοσιονομική γραμμή ή πιλωτικές δράσεις. Ε, αναγνωρίσαμε την σημασία τους και τα συμπεριλάβαμε στους βασικούς α, τίτλους. Εγώ μπορώ να το συζητήσω με τον εισηγητή. Είναι σημαντικό να έχουμε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε τις ιδέες μας ε, και να δούμε λεπτομερώς τα νούμερα. Τέλος, τον ευχαριστώ για τα σχόλιά του, για τις ε, διοικητικές πιστώσεις. Πιστεύουμε ότι στο σχέδιο προϋπολογισμού οι προτάσεις που έχουν ε, γίνει είναι ρεαλιστικές και συνάδουν με την αύξηση που υπάρχει σε άλλες πιστώσεις. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού θέλουν να πούν δύο λόγια. Κυρία Πρόεδρε, είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού. Ε, να συμπληρώσω τις ε, δηλώσεις του συναδέλφου από την Κομισιόν, να κάνω κι εγώ κάποιες ε, παρατηρήσεις για τη χρηματοδότηση για την, ε, για την κλιματική αλλαγή. Η πρόταση που υπάρχει επιτάπητο σήμερα για τον προϋπολογισμό 2011 είναι μια πρόταση συμπληρωματική, επιπρόσθετη. Έτσι, συμπληρωματική. Και πέρυσι ήταν ε, συμπληρωματική και φέτος είναι επιπρόσθετη. Και του χρόνου ε, στο δημοσιονομικό προγραμματισμό, όχι στο προϋπολογισμό, το προτείνουμε του χρόνου. Έτσι, στον προγραμματισμό προτείνουμε αυτό το επιστέγασμα. 50 ε, εκατομμύρια ε, σε σχέση με τα 7,2 δις ε, για τρία χρόνια. λίγα λεφτά, αλλά είναι μια συνεισφορά για την επιστηστική ασφάλεια που αποφασίστηκε, αυτά που είπε ο εισηγητής σας, το ίδιο σχόλιο με του συναδέλφου μου είναι ε, μια συνιστόσα της DCI ε, που αυξήθηκε κατά 31% ανάμεσα στο 2007 και το 2013. Δηλαδή είναι το, η συνιστόσα που αυξήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Πρόκειται για ποσά DCI και υπό ποσά τα οποία αυξάνονται και που καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου προγραμματισμού αυξάνονται. Ε, χάρη στις παρεμβάσεις της Δημοσιονομικής Αρχής, δηλαδή εσάς και του Συμβουλίου. Σε ό,τι αφορά τώρα την κατάσταση του τίτλου 4, που χρόνια τώρα υποπρικοδοτείται και έχει έλλειμμα κονδυλίων, αν αυτό είναι από τα συμπεράσματα της Επιτροπής στην έκθεση που αναφέρθηκε και που βγαίνει παράλληλα με το σχέδιο προϋπολογισμού του 2011, στο τέλος αυτού του εγγράφου ε, ουσιαστικά ξεκινάει η συζήτηση για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού φέτος. Τώρα θα ξεκινήσει, γιατί η Κομισιόν καθυστέρησε κατά 6 μήνες την παρουσίασή της. Και λέει ότι για τις σημαντικές ανάγκες, πολύ συγκεκριμένες και εστιασμένες και οριοθετημένες, μπορούμε να αλλάξουμε το νοτοτόριο. Και αναφέρουμε ως παράδειγμα στο έγγραφο της Κομισιόν που δόθηκε σήμερα το πρωί την προσπάθεια για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Για ε, το τελευταίο σημείο που αφορά, όπως που αφορά τις διοικητικές δαπάνες, τις δαπάνες για τη διοικητική στήριξη που ανέφερε και ο κ. Πάντιγκτον, η Κομισιόν βασίστηκε στην απόφαση της Δημοσιονομικής Αρχής που ελήφθη πέρυσι. Ε, επικυρώσαμε αυτή την απόφαση και αυξήσαμε τις δαπάνες αυτές ε, με προσαρμοσμένο τρόπο ανάλογα με την αύξηση των ποσών γενικότερα. Ε, αυτό συνάδει με την πολιτική απόφαση του Κοινοβουλίου πέρυσι και με την αύξηση γενικότερα των πιστώσεων και ποσών. Ε, σε αυτόν τον τομέα, σε άλλους τομείς, σε άλλες πολιτικές, δηλαδή την διεύρυνση, τα ποσά που προβλέπονται για διοικητικά θέματα είναι πολύ λιγότερα. Είναι τα μισά ή το 1 τρίτο ε, από ό,τι προβλέπουμε για τον DCI. Ε, είναι τελείως δικαιολογημένο αυτό. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τα ίδια πράγματα, ας πούμε, στην Ασία, στην Αφρική ή στην Τουρκία και στην Κροατία. Η Κομισιόν θέλει να υπάρχει σωστή ισορροπία και αυτό είναι το παράδειγμα της σωστής ισορροπίας. Αυτά και είμαστε στη διάθεση του εισηγητή για να συμπληρώσουμε τις παρατηρήσεις μας και γραπτός πάνω σε αυτή την εξαιρετική του έκθεση. Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, τώρα τα μέλη της Επιτροπής μας. Ε, υπάρχουν σχόλια? Ο κύριος Γκόρεντς. Ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση για τα 2,4 δις. Επένδυση δηλαδή για τα προγράμματα για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών σε αναπτυσσόμενες χώρες. Νομίζω ότι όλοι δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε. Ποια είναι η χρηματοδοτική τεχνική του μέτρου αυτού. θα τα συλλέξει η Επιτροπή τα κονδύλια και θα χρηματοδοτηθεί δηλαδή αυτός ο πόρος από τα κράτη-μελή. Αυτό ισχύει όντω. Αν ναι, έχω και ε, επερωτήσεις για τα επιπρόσθετα κονδύλια. Να, ας ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις μαζί ίσως, λέει η Πρόεδρος. Όχι. Απάντηση. Κύριε Γκέρενς, Ναι, στον ε, τωρινό δημοσιονομικό κανονισμό δεν έχουμε μέσα για να συλλέγουμε πόρους από τα κράτη-μέλη. Τα 2,4 είναι πιστός ανάληψη υποχρεώσεων μάλλον ε, ανάληψη υποχρεώσεων και από πλευρά τη Επιτροπή και από πλευρά των ε, κρατών μελών. Αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα περάσουν όλα τα λεφτά μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν θα τα συλλέξει η Επιτροπή δηλαδή. Επερώτηση. Νομίζω πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για τα 2,4 δισεκατομμύρια. Συμφωνώ ε, με την εισήγηση ότι πρέπει να πρόκειται για επιπρόσθετα κονδύλια. Το έχουμε πει επανειλημμένως. Για να ξεφύγουμε από την παγίδα του επαναχαρακτηρισμού της βοήθειας, της επαναταξινόμησης της βοήθειας, ε, η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει το καθήκον της και Παρεπιπτόντως δεν έχω κάνει καμία αμφιβολία εγώ. Φυσικά τα ε, λεφτά που θα πάρετε από τα κράτη-μέλη θα είναι τα κονδύλια. Δεν ρώτησα αυτό. Τα κονδύλια που έρχονται από τα κράτη-μέλη θα τα έχετε πάρει από ένα κομμάτι του προϋπολογισμού που ήδη ε, αφιερώνεται σε άλλους αναπτυξιακούς στόχους γιατί τότε μιλάμε για επαναχαρακτηρισμό της βοήθειας και δεν πρόκειται για επιπρόσθετα κονδύλια και βάσει της ε, συνθήκης της Λισαβόνας ε, τονίστηκε ανάγκη να υπάρχει συνοχή της πολιτικής σε επίπεδο ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών. Γι' αυτό έχει τόση μεγάλη σημασία αυτή η λεπτομέρεια. Στην Κοπενχάη και γι' αυτό επιμένω η Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησε σαφέστατα σχετικά με το αν είναι επιπρόσθετα κονδύλια με ένα ίξις αφήξη στυλ. Ε, πρέπει να μάθουμε τι, τι ισχύει εν πάση περιπτώσει και να μην μας λένε ιστορίες για γρίους. Ευχαριστούμε ε, κύριε Γκόρες. Ο κύριος Τυρόλιαν. Euh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ παρά να συγχαρώ τον εισηγητή μας για την παγρύπνησή του που υπογράμμισε πραγματικά ε, τι εστί ε, εργαλείο χρηματοδότησης ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα κάνει μια πρόταση τροποποίησης του μέσου αυτού για να χρηματοδοτεί ε, μια τετραετία με 180 εκατομμύρια ευρώ ε, τα συνοδευτικά μέτρα για τους παραγωγούς μπανάνα ΑΚΕ όπως συμφώνησαν στον ΠΟΕ το Δεκέμβριο που μας πέρασε. Όμως θα πρέπει να υποστηρίξουμε ε, με επιπλέον πόρους τις νέες αλλαγές και η πρόταση αυτή είναι απαράδεκτη. Αυτοί προτείνουν να πάρουν από το ε, μέσο της αναπτυξιακής βοήθειας χρήματα που προορίζονται για την υγεία, για την ανάπτυξη των χωρών που έχουν προβλήματα με την οικονομική κρίση για να χρηματοδοτηθεί η μπανάνα. 75 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ το 2010 θα πάρει από αυτό το μέσο DCI. Ε. Ή 18,3 μόλις από το μέσο ευελιξίας αυτό το μέσο όμως έχει πολλά χρήματα και φρέσκο χρήμα, πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε ε, να αντλήσει από εκεί περισσότερα χρήματα παρά να αποψηλώνει ε, γραμμές του προϋπολογισμού που είναι τόσο σημαντικές για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τη στιγμή που ξέρουμε ότι θα είναι σχεδόν αδύνατο να πετύχουμε όλους τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας μέσα σε πέντε χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνει ένα πολύ κακό μήνυμα και θα επιθυμούσαν να μας απαντήσει τα ερωτήματά μας και να ε, μας διευκρινίσετε την οδήγησε να αποφασίσει ε, αυτά που αποφάσισε. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στη δημοσιονομική διαδικασία για να αποφύγουμε αυτό το νέο γδίσιμο του ε, μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας. Ευχαριστώ. Well, Τώρα ο κύριος Γκουτική ρώτησε ναι, δεν υπάρχει κανένα άλλο συνάδελφο που έχει στήσει το λόγο προηγουμένω. Ε, ε Αλλιώ να περιμένω. Κανεί άλλο δεν θέλει, τότε να μιλήσω εγώ. Ωραία. Και αυτό που είπα προηγουμένω συνδέεται με τούτο εδώ. Δεν παίρνουμε από τον ένα, με τον ένα χέρι να το δώσουμε στον άλλον. Ε, δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί πάντα να υπερασπίζεται τις αντιφάσεις των κρατών μελών. Το καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να ακούσω και το Συμβούλιο, γιατί είναι θέμα Συμβουλίου. Δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απολογείται εδώ για το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δίνει την εντολή για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Άρα το Συμβούλιο θα πρέπει να λογοδοτήσει στο Κοινοβούλιο μα Οφείλει απαντήσει από αυτό. Γιατί εάν θέλουμε να βρούμε ε, μια λύση θετική στο πρόβλημα της μπανάνας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τόσο στη δεν ξέρω, το Συμβούλιο θέλει να μιλήσει από αυτό. Αλλιώς δεν θα έχουμε ποτέ συνάφεια και συνοχή σε αυτά που λέμε. Και ποιος ε, ε, τώρα θα καλούμαστε να μαντεύουμε τι σκέφτεται το Συμβούλιο. Θέλει κανείς να απαντήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει πρόεδρος. Council. Το Συμβούλιο. Ο εισηγητής ίσως. Ah, Α, η Κομισιόν. Excuse me. Euh, Ευχαριστώ για την προσθετικότητα. Ε, δεν μπορεί τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφανθεί για τις εξαγγελίες των κρατών μελών ε, στην Κοπενχάγη αφού δεν έχουν ακόμη πραγματοθεί στο Συμβούλιο. Ε, συνεχίζω τις συζητήσεις για αυτά τα σημεία. Για τα 2,4 δις που συμπεριλαμβάνουν και την υπόσχεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, δεν μπορούμε τώρα και εδώ να ε, εκφέρουμε άποψη. Ελπίζω αργότερα. Τα κράτη-μέλη, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τοποθετηθούν. Αυτό που είπε ο κύριος Κόρενς, ε, κατά πάσα πιθανότητα έχει σημασία για την Επιτροπή σας. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα δεν είναι σε θέση να αποφανθεί για τα 150 εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, εντάξει είναι χαμηλό όπως εφόσον μιλάμε για 7,2 δις για μια τριετή περίοδο. Βγάλαμε όμως φρέσκα λεφτά, θα βγάλουμε φρέσκα λεφτά. Και γι' αυτό στην απάντηση που σα στείλαμε, μιλάμε για την προσθετικότητα σε σχέση με τον νοσιακό προπολογισμό. Είναι φρέσκα τα κονδύλια. Είναι ένα κομμάτι τη απάντηση που δίνουμε. Μπορεί να μην έχει αρκετό βάρος, αλλά αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα. Ε, για το μέτρο για την μπανάνα. Πρώτον, κατά 50% το μέτρο αυτό θα έχει και αυτό νέα κονδύλια, φρέσκα κονδύλια, έτσι, κατά το ίμιση χρηματοδοτείται από νέα κονδύλια. Για τα υπόλοιπα, για να χρησιμοποιήσουμε το μέσο ευελιξίας που έχει μέσα η διαθεσμική συμφωνία, οφείλει, οφείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάει να ψάξει χρηματοδο... Ε, ε, θύλακες όπου υπάρχει υποαπορρόφηση κονδυλίων. Και άρα μέσα στα διάφορα ε, μέσα, όχι μόνο στο DCI, να βρει τους θύλακες ε, για το μελλοντικό προγραμματισμό. Πού υπάρχουν αδυναμίες για το DCI, το DCI αντιστοιχεί μόνο σε 10-13% του ποσού. Δεν αποψηλώνουμε λοιπόν ε, το ένα για να ντύσουμε το άλλο. Πρόκειται για ανάγκες μελλοντικού προγραμματισμού. Το κονδύλι της ΙΑΗ γενικά και στη, σε λεπτομέρεια συνεχώς αυξάνεται. Γιατί αυτό θέλησαν νομοθετικές αρχές και για την επόμενη περίοδο. Αλλά πέραν αυτού έχουμε και επιπρόσθετα 400 εκατομμύρια, ε, δηλαδή 400 ε, εκατομμύρια που έχουν προσθεθεί από την αρχή της προγραμματικής περίοδου. Αυτά. Ε, τώρα για τη γνώμη του Συμβουλίου, να απαντήσει το Συμβούλιο, έτσι, άμα μπορεί είναι στην πρώτη συζήτηση προς το παρόν. Αλλά ε, κύριε βουλευτές, ε, νομίζω ότι ε, καταλαβαίνετε πως δεν θα αρέσει στο Συμβούλιο αυτή η αλλαγή στο χρηματοδοτικό μέσο. Δεν χρειάστηκε για γυάλινη σφαίρα για να το προβλέψετε αυτό. Ελπίζουμε να τύχει θετική υποδοχή η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντω, η ίδια η Επιτροπή δεν μπορεί να κινητοποιήσει το μέσο ευελιξία αν πρώτα δεν βρει ε, θύλακε υποαπορρόφηση ε, για να ε, αναδιαθέσει τα κονδύλια. Θέτουμε πρώτον ευθυνότητα το Συμβούλιο. Έτσι. Καταλαβαίνω ότι έχει διαφορετικέ ανησυχίε το Συμβούλιο, αλλά το καθήκον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό είναι, γιατί αυτό μα ζητάει η διαθεσμική συμφωνία. Αυτά τα σχόλια έχω να κάνω για τα δύο ζητήματα που πήγαιναν οι βουλευτές. Γκέρεν. και άλλη μια επιπρόσθετη ερώτηση. Μόλις είπατε ότι το 50% των χρημάτων είναι νέο χρήμα σε αυτές τις δράσεις. Στο κείμενο το οποίο συνοδεύει τον προϋπολογισμό, πώς τον λέτε στα γαλλικά, Υπάρχουν 75 εκατομμύρια το 2010 για τη δράση για τις μπανάνες, εκ των οποίων 18,3 εκατομμύρια προέρχονται από το FLEX, το εργαλείο για την ευελιξία. Και το υπόλοιπο είναι το υπόλοιπο. Αν πάρουμε ένα εκατομμύριο από εδώ και ένα εκατομμύριο από εκεί, αυτό τι είναι, είναι χρήματα που τα παίρνουμε από εδώ και τα χρησιμοποιούμε εκεί. Πού είναι αυτά τα 50 φρέσκα κονδύλια. 18 ε, στα 75 εκατομμύρια. Πού είναι τα νέα χρήματα, εν περιπτώσει, το 50% που είναι νέο, φρέσκο χρήμα. Εξηγήστε μου σας παρακαλώ, Κομισιόν, δεν το βλέπω. Χωρίς να θέλω να παρατείνω τη συζήτηση για αυτό το θέμα, το δικό μου ε, σχόλιο αφορούσε τα 190 εκατομμύρια για την περίοδο. Σε αυτά τα 190, το 50% είναι νέο χρήμα. Η ευελιξία, το, το εργαλείο για την ευελιξία λοιπόν προβλέπει νέα κονδύλια. 190 φέτος για την ε, περίοδο, για τη μοναδική περίοδο που προτείνουμε το εργαλείο για την ευελιξία, γιατί για τα επόμενα χρόνια δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε. Ε, κατά τα άλλα τα νούμερα είναι αυτά που είπατε. Εγώ μιλάω για τη χρηματοδότηση 190 με τα 190 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα είναι ευελιξία ή ε, μετατόπιση κονδυλίων. Όχι μόνο DCI, έτσι. Μπορούμε να σας δείξουμε και τα νούμερα, κύριε Μπέρμαν, για να τα καταλάβετε. Thank you and Mr. Ευχαριστώ, κύριε Γκέρενς. Και ο κύριος Γκέρενς, μάλλον. Λοιπόν, δεν θέλω τώρα να κάνω διελκυστίνδα με την Κομισιόν. Μιλάτε για 150 εκατομμύρια ευρώ, έτσι για να διευκολυνθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Μπράβο. Ωραία. Το θέμα είναι, οι άλλοι θα ακολουθήσουν. Ε, τα κράτη-μέλη δηλαδή θα δώσουν επιπρόσθετα χρήματα. Έχουμε εδώ μια ξεκάθαρη θέση. Θα πρέπει να είναι επιπρόσθετα χρήματα. Γιατί αλλιώς διηγούμεθα παραμύθια στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, για αυτή τη νέα συμφωνία για την κλιματική αλλαγή. Εγώ προτείνω στον εισηγητή να στείλει μια επιστολή εξ ονόματο της Επιτροπής μας στο Συμβούλιο για να διευκρινιστεί αυτό το σημείο. Γιατί και η, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η δική μας Επιτροπή θέλουμε να ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα. Στο προήμιο της επιστολής του θα μπορούσε να πει ότι και τα κράτη-μέλη καλό θα ήταν να δεσμευθούν να αυξήσουν την αναπτυξιακή βοήθεια κάθε χρόνο. Ε, και θα πρέπει να υπάρχει και ένα περιθώριο για φρέσκο χρήμα, επιπρόσθετα κονδύλια. Θα πρέπει νομίζω να ξεκαθαριστεί αλλιώ αυτό, γιατί αλλιώ χάνουμε το χρόνο μα. Το καλύτερο είναι να αντιδράσει το Συμβούλιο. Ε, και εσεί στην ίδια θέση είσαστε κομισιόν με εμά. Ε, είμαστε και οι δύο σε θέση αναμονή ουσιαστικά. Εγώ αυτό προτείνω να κάνετε. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο κ. Μπέρμαν ω εισηγητή, να ολοκληρώσει. Όχι, Πρόεδρε. Ξεκαθαρίσαμε ότι επιμένουμε ε, στο σημείο της ε, προσθετικότητας για όλα τα μέτρα που συνδέονται με το κλίμα και με τα υπόλοιπα θέματα ε, και που δεν συνδέονται άμεσα με την ελάφρυνση της φτώχειας. Νομίζω ότι ένα από τα προνόμια του να ε, συμμετέχει κανείς σε αυτήν την επιτροπή να, να, να υπενθυμίζει τέτοιες θέσεις. Υπενθυμίζω uh, η ημερομηνία για τις προθεσμίες είναι 3 Μαΐου. Τώρα πάμε στο σημείο 15 και 16 της ημερήσιας διάταξης μαζί η θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη διάσκεψη κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Τορόντο 26-27 Ιουνίου 2010 για την ανάκαμψη και τις νέες και τη νέα αρχή, το G20, θα εστιάσει στην ανάκαμψη από την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι προηγούμενες συνοδικορυφείς G20 και θα εξετάσει πώς θα τεθούν τα θεμέλια για μια βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη. Υπάρχουν τρία βασικά θέματα που θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφή. Αναθεώρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, προγράμματα κινήτρων και παγκόσμιο εμπόριο και, ανα, και ανάπτυξη. Αυτά τα τρία θέματα έχουν άμεση επίπτωση στι αναπτυσσόμενε χώρε, γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε δύο πράγματα. Καταρχά, ε, να στείλουμε μια επιστολή στον Καναδό Πρωθυπουργό Χάρπερ για να ζητήσει από τη Σύνοδο Κορυφή ε, του G20 να ενθαρρύνει του ηγέτε του κόσμου να λάβουν δράσει για να προωθήσουν τι προσπάθειε εξάλληψη τη φτώχεια και την ε, προώθηση τη χρηματοπιστωτική ανάπτυξη, την καταπολέμηση των παράνομων κεφαλαιακών ροών ε, που φεύγουν από τις, ε, από τις αναπτυγμένες χώρες. Έχουμε το κείμενο αυτής της επιστολής ε, και το έχετε και εσείς στο φάκελό σας. Επίσης θα ακολουθήσει θα μια υποβολή μιας προφορικής ερώτησης υπό το άρθρο 115 του Συντερικού κανονισμού και θα κάνουμε αυτή τη δήλωση στην Ολομέλεια οι πολιτικές ομάδες ε, ζήτησαν και η Γραμματεία έχει προετοιμάσει το σχέδιο αυτής της προφορικής ερώτησης ε, της Επιτροπής μας, ε, καθώς και το ψήφισμα. Αυτά τα κείμενα έχουν διανεμηθεί και έχουν διδράσει πολιτικές ομάδες. Σημειώστε ότι η προφορική ερώτηση και το σχέδιο ψηφίσματος προβλέπονται για την επόμενη συζήτηση της 10ης Μαΐου. Τώρα θα ζητήσω από την Επιτροπή να σχολιάσει και την ερώτηση και το σχέδιο ψηφίσματος και να μας ενημερώσει για τη θέση της για τη συνάντηση του G20. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ουσιαστικά ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εν συντομία θα ήθελε να σχολιάσει τις συζητήσεις που έγιναν πρόσφατα στη G20 για το θέμα αυτό. Ξέρετε ότι παρουσιάστηκε σε εκείνη την διάσκεψη ε, με ένα σχέδιο έκθεσης, ενδιάμεση έκθεση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, το οποίο δεν κοινοποιήθηκε στον τύπο. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι κάποια από τα σημεία της έκθεσης δεν συνάδουν με τις ε, τεχνικές συστάσεις του πρόσφατου εγγράφου εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό δείχνει τις δυσκολίες ε, που υπάρχουν σχετικά με την εισαγωγή ε, φόρων σε, σύγκριση με τη χρήση ε, άλλων εργαλείων. Το πρόβλημα με το, τη φορολόγηση των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μέσα στην έκθεση και στο έγγραφο εργασίας μας είναι ότι ε, όντως μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική συλλογή εσόδων αλλά ε, το θέμα είναι κατά πόσο θα κοινοτομήσουμε με αυτόν τον τρόπο και πού θα, πώς θα ανακατανεμηθούν αυτά τα έσοδα. Επίσης, ε, το πώς θα επηρεάσει αυτό τη σταθερότητα του ισολογισμού κάποιων επιχειρήσεων. Ναι, μεν συλλέγουμε έσοδα, αλλά ε, φορολογώντας τις ε, χρηματοπιστωτικές ε, συναλλαγές ε, δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Πρέπει να αποφασίσει κανείς σε ποια μέσα θα το εφαρμόσετε, σε ομόλογα, σε παράγωγα, σε, γενικά σε χρεόγραφα είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τον αντίκτυπο και μπορεί να επιβαρύνει δυσανάλογα πολύ κάποια χρηματοπιστωτικά μέσα και το ε, συλλεχθέν εισόδημα την εστιάζεται σε κάποιες χώρες που έχουν μεγάλα ε, χρηματοπιστωτικά κέντρα και παίρνουν ανάλογα μεγάλο κομμάτι αυτών των εσόδων, οπότε η κατανομή των βαρών μπορεί να δημιουργήσει επίσης πρόβλημα. Η ανάλυση της Επιτροπής επίσης σημειώνει τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με το ότι μπορεί να είναι ασύμβατες αυτές οι διάταξει ε, σχετικά με το άρθρο 11 ε, τη Συμφωνία ε, Γκάτσε αλλά και με τον σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών μέσων. Κάποιες αναδυόμενες αγορές δεν υποστήριξαν αυτή την πρόταση στις, από από τη ΣΥΠΑ υποστηρίχθηκε ε, το τέλος για τη σταθερότητα των ισολογισμών των επιχειρήσεων, ε, αλλά δεν υπήρξε ε, θετική υποδοχή για αυτού του είδους τη φορολόγηση. Στην G20 Αναμενόταν αυτή η τελική έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά επίση ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υπήρχε ε, ευρεία συνένεση, τουλάχιστον όχι τόσο ευρεία όσο θα περίμενε κανεί, το οποίο σημαίνει επίση ότι μπορεί να είναι τελικά πιο δύσκολο να εφαρμοστεί ευρύτατα ένα τέτοιο μέσο φορολογικό. Οπότε το σχετικό πλεονέκτημα όπως το τέλος σταθερότητας που δεν χρειάζεται τόσο ευρύ, ευρύ διεθνή συντονισμό παρότι θα χρησιμεύω συντονισμός για τέτοια μέσα. Ε, αυτό λοιπόν πρέπει να τονιστεί. Άρα η Επιτροπή σε εκείνη τη συνεδρία τόνισε τη σημασία του παγκοσμίου συντονισμού, τη ε, συμφωνία για κάποιε βασικέ αρχέ ε, για τέτοια μέσα. Όχι απόλυτα μειομορφία, δεν επιδιώκουμε αυτό, αλλά τουλάχιστον να συμφωνήσουμε για κάποιε γενικέ αρχέ, ε, ούτω ώστε να μειώσουμε τι τρευλώσει του ανταγωνισμού και τι κανονιστικέ αυθαιρεσίε. Πάντως θεωρούμε ότι ήταν χρήσιμη αυτή η έκθεση. Ευχαριστούμε. Θέλει κάποιο να σχολιάσει αυτό το σχέδιο ερώτηση ή το σχέδιο ψηφίσματος, ο κύριος Γκερέιρο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αλλά εξαφανίζεται η Πρόεδρος. πρέπει να πω κύριε Πρόεδρε στο φτερό αλλάζουν οι πρόεδροι. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό το θέμα που μου φαίνεται αρκετά σημαντικό. Αρχίζω από το πλαίσιο που μας επιτρέπει να συζητούμε σήμερα για αυτό το θέμα. Πιθανότατα πριν από τρία χρόνια να μην γινόταν αυτή η συζήτηση ούτε καν στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Και δεν μιλάω καθόλου για άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Γιατί συζητούμε σήμερα αυτό το θέμα. Διότι ως απόρρια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και του αντικτύπου που είχε παντού, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι θα ήταν σκόπιμο σε πρώτο λόγο να ε, ρυθμίσουμε τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, τις οποίες οφείλεται η κρίση, και σε δεύτερο λόγο να βρούμε νέες πηγές χρηματοδότησης για την καταπολέμηση της ένδυας και τη βοήθεια των αναπτυσσομένων ε, κρατών. Στην αρχή, το G20 ε, είχε την βίκονους σε αυτές τις ε, σκέψεις μας. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και όσο για μερικές χώρες η κρίση περνάει και απομακρύνεται και μένει πίσω, η όθηση για να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση δεν είναι ημιούμενη και η απροθυμία μεγαλών. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο ή παράθυρο ευκαιρίας όπως ονομάζεται για να οθήσουμε το G20 ή άλλα διεθνή χρηματοοικονομικά ιδρύματα να πάρουν μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Και θα πρέπει να ε, αξιοποιήσουμε την επόμενη συνεδρίαση, διότι επιπλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο στο Συμβούλιο Κορυφής θα έχουν σημείο στην ημερήσια διάταξη, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δηλαδή, για την ανάπτυξη. Οπότε έχουμε τώρα 15 μέρες που εκτός του παγκοσμίου ε, κυπέλου ποδοσφαίρου ε, φιλοδοξεί η χώρα μου να το πάρει, έτσι. Α είμαστε όμω συγκρατημένοι στην ισοδοξία ε, μα, γιατί ποιο ξέρει. Όχι, λέει ο κύριο Κάσμαν, εμεί θα το πάρουμε. Καλά. 15 ε, μέρες ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνεδριάζει και θα συζητάει και για την ανάπτυξη. Και το G20 επίσης στην αρχή θα συζητήσει πολλά και διάφορα άλλα θέματα, αλλά είναι ευκαιρία να βάλει στη μερίσια διάταξή του και αυτά τα θέματα της ανάπτυξης. Και εδώ και στην ερώτηση λοιπόν, αλλά και στο ψήφισμα έχουμε μια σειρά αποζητήματα τα οποία είναι θετικά όλα για να προχωρήσουμε, σε περίπτωση που θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη. Ε, ε, κατά πολέμηση της φοροδιαφυγής, πολέμηση των φορολογικών παραδείσων, πολέμηση της τάσης που έχουν οι εταιρείε να κρύβουν τα κέρδη τους, ε, ανάλογα με τις χώρες τις οποίες δραστηριοποιούνται. Και τέλος, και ένα τέλος για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Στο G20 τώρα διαφαίνεται μια τάση και στις χώρες γενικά ε, το τέλος αυτό να το χρησιμοποιήσουν για να σταθεροποιήσουν ε, το τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή να πάρουν τα λεφτά από τις χρηματικές συναλλαγές για να εξασφαλίσουν το υπάρχον χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εμείς δεν ζητάμε κάτι τέτοιο, ούτε αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Ε, τι ζητάμε, αυτούς τους πόρους, τους οικονομικούς που θα αποκομίσουν ενδεχομένω από το τέλος αυτό, θα πρέπει να τους, στείλουμε, να τους διοχετεύσουμε στην καταπολέμηση της φτώχειας και της του αποκλεισμού, συγγνώμη. Όπω, ε, μόλις είπε ο πρόσωπος Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι συγκεκριμένη θέση του G20. Μερικέ χώρες είναι ε, περισσότερο υπέρ από κάποιε άλλες ε, του τέλου αυτού. Και ε, μέσα και στους υπέρ πάλι δεν ξέρουν ακριβώ τι φόρος θα αυτό τι τέλος και πώ θα οργανωθεί. Αυτό που εμεί τώρα όμω προσπαθούμε να στοιχειοθετήσουμε με την έκθεση αυτή, με την ερώτηση μάλλον και το ψήφισμα και τη συζήτηση είναι Ποια είναι η ηθική και πολιτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη συζήτηση. Πέρα δηλαδή από το τεχνικό αποτέλεσμα που ουσιαστικά ενδεχομένω να προκύψει και να τεθεί σε λειτουργία μετά από έγκριση κάποιου είδους φόρου ή τέλους, αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι αν θα εξακολουθούμε να είμαστε στην πρωτοπορία εκείνων που ζητούν τέτοιες μεταρρυθμίσεις, αν θα συνεχίσουμε να είμαστε, πώς να το πω, ένα παράδειγμα προς μίμηση ε, από άλλες πλούσιες χώρες ή δυνάμεις του κόσμου. Ή αντιθέτως αν παραδεχτούμε ότι ε, πέρασε η κρίση στο μεγαλύτερο βαθμό και συμβαζόμαστε με τη θέση που είχαμε το 2007 και επιστρέφουμε σε αυτή. Και όπως είπε προηγουμένως και ο Τάις Μπέρμαν, και εγώ είμαι περήφανο που ανήκω σε τούτη εδώ την Επιτροπή και αγωνίζομαι όχι για να επιστρέψουμε στο 2007, αλλά να κάνουμε μεταρρυθμίσεις για το 2010 κτλ. Ευχαριστώ. So, Mrs. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για αυτό το ψήφισμα, για το G20. Καταρχάς, προσοχή. Νομίζω ότι το 2010 ψηφίσαμε στο Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα για το θέμα των φόρων. Για μας, λοιπόν, θέλουμε να προτείνουμε κάτι καινούριο, να μην επαναλάβουμε τα ίδια. Ένα νέο ψήφισμα έχει νόημα κατά την άποψή μου μόνο αν διευρύνουμε το ψήφισμα που θα εξετάσουμε και περιλάβουμε θέματα ε, διαφάνειας και δημοσιονομικής διαχείρισης. Ο κ. Γκερέρο μίλησε για το πλαίσιο. Ε, θέλω να επανέλθω στην προηγούμενη συνοκορυφή του Πίτσπουργκ που κατά την άποψή μας δεν ήταν ικανοποιητική. Αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε με το νέο ψήφισμα είναι να αναπτύξουμε μηχανισμούς κυρώσεων και να είμαστε πολύ πιο ρητοί και ξεκάθαροι για το θέμα του τραπεζικού απορρίτου. Ο κύριος Γκερέρο μίλησε για το αν θα παραμείνουμε πρωτοπόροι ε, στα θέματα των φορολογικών παραδείσων. Εγώ προτείνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπερασπιστεί στη διεθνή σκηνή ε, αυτά που κάνει στο εσωτερικό της. Δηλαδή μια αυτόματη ε, ενημέρωση, ε, αυτόματη, επαναλαμβάνω, για όλα τα τραπεζικά δεδομένα. Θέλω να κλείσω με δύο παρατηρήσεις. Η θέση για τους φορολογικούς παραδείσους δεν είναι μόνο ηθικής διάστασης ιδεοντολογικής διάσταση, Ε, θέλω να υπενθυμίσω ότι η φορολογική παράδειση δημιουργούν και αθέμητο ανταγωνισμό σε οικονομικό επίπεδο και μία σκέψη που θα πρέπει να μας απασχολήσει για το G20 που θα γίνει τώρα, για τη συνοκορυφή στην καινούρια. Είναι το θέμα της, νομιτο... της νομιμότητας. Τι νομιμότητα υπάρχει όταν αποκλείουμε 172 χώρες. Και τελικά, ο ρόλος μας δεν είναι να προωθήσουμε ε, με έδρα τον ΟΗΕ. Να συμβαίνουν δηλαδή αυτές οι συζητήσεις κυρίως και βασικά στο εσωτερικό του ΟΗΕ. Κύριος Κάσμαν, ε, ζητώ συγγνώμη τον εκπρόσωπο της Κομισιόν που δεν ήμουν ε, εδώ ε, όταν έκανα την παρουσίαση. Ε, παίρνω το λόγο γιατί συζητάμε από ό,τι κατάλαβα καλά το σημείο 15 και 16 μαζί. Βασικά θα τοποθετηθώ για το σημείο 16, αλλά βέβαια είναι αλληλένδετα. Ε, η προφορική ερώτηση που θα κλείσει το ψήφισμα για τη θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τη σύνομα κορυφής του G20 και κυρίως για το φόρο ε, για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Ο πρόεδρος Παρόζο, αν θυμάμαι καλά, δήλωσε το Δεκέμβριο ότι θεωρούσε ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα αυτή η ιδέα του φόρου. Και το Κοινοβούλιο ήδη έχει λάβει θέση για αυτό το θέμα. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι έγιναν συζητήσεις ε, και στην Επιτροπή για ένα φορολογικό τέλος χρηματο χρηματοπιστωτικό, αν θέλετε τέλος, 0,09% αν δεν απατώμε. Αυτό το νούμερο ακούστηκε. Και εγώ το αναφέρα και στην δική μου έκθεση για τους στόχους της χιλιετίας. Αλλά δεν αναφέρω πια ποσοστό, γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τον G20 και άλλους να είναι πολύ πιο φιλόδοξοι και να μιλήσουν για ποσοστά ανώτερα και να αναγνωρίσουμε ότι αυτό που ζητάμε δεν είναι απλώς ένα τέλος για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη και σε άλλους να ε, σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους για το 0,7 της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά για να κάνουν κάτι παραπάνω. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα συμφωνήσουμε, πώς θα φτάσουμε σε μια συμπεφωνημένη θέση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, στο επόμενο summit ε, για αυτό το φόρο για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Υπάρχει σχέδιο για να εξασφαλίσουμε ότι τα έσοδα θα θεωρηθούν πρόσθετη χρηματοδότηση. Πρόσθετη, το υπογραμμίζω. Και πώς θα υποστηρίξουμε την ιδέα ότι αυτή η επιπρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κατεπίγουσες ανάγκες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κυρίως, όπως είπαμε και πριν, ε, μετριασμού των κλιματικών αλλαγών, για τέτοια θέματα. Αυτέ είναι οι αρχικέ μου σκέψει και ζητώ συγγνώμη ξανά που δεν ήμουν εδώ όταν εκπρόσωπο τη Κομισιόν έκανε την παρουσίασή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κάσμαν. Θέλει να απαντήσει η Επιτροπή. Ε, είναι δύσκολη η συζήτηση για τα διάφορα εναλλακτικά σενάρια, αλλά υπάρχει ευρεία συνένεση ότι χρειάζεται ε, ένας τρόπος για να μεριμνήσουμε ώστε ο χρηματοπιστωτικός ε, τομέας να αναλάβει το κόστος που επέβαλε στη ολόκληρη την κοινωνία και στους δημόσιους προϋπολογισμούς. Διάφορες κυβερνήσεις, όχι μόνο στην Ευρώπη, ε, τείνουν να συμφωνήσουν για ένα είδος τέλους ε, σταθερότητας παρά ε, για ένα φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Το σημαντικό είναι να υπάρξει συνένεση για ένα από τα σενάρια. Όπως είπε ο Ισπανός βουλευτής, μπορεί να παρεπεράσει, να κλείσει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που ανοίγει τώρα. Αν δεν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα συνδυασμό των δύο μέσων. Ε, δεν χρειάζεται να εστιάζουμε μόνο σε ένα μέσο και μπορούμε, αν αρχίσει να διαφαίνεται μια συνένεση, να τη χρησιμοποιήσουμε. Εάν στη G20, 20 σας είπα ότι δεν υπήρξε ε, υποστήριξη, ευρεία συνένεση για αυτό το φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, οπότε μπορούμε να βασιστούμε σε άλλες προτάσεις ε, για να έχουμε έσοδα, για να ε, πληρώσει το τίμημα που το αναλογεί ο χρηματοπιστωτικό τομέα. Και ένα άλλο ζήτημα είναι πώ θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια. Το έγγραφο εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν ε, αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Ε, δηλαδή η διάθεση αυτών των κονδυλίων, η δεσμευσή τους είναι ένα λεπτό πολιτικό ζήτημα, αλλά είναι σαφές ότι αν από το χρηματοπιστωτικό ή το τραπεζικό σύστημα λαμβάνουμε περισσότερα κονδύλια τότε θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ε, αναπτυξιακέ δράσεις και δράσεις ε, για την αντιμετώπιση των ε, κλιματικών αλλαγών. Ευχαριστούμε. Περάτησε ο κύριο Κάσμαν. Ευχαριστώ. Συμφωνία από το τραπεζικό σύστημα. δηλαδή πότε ψήφισαν οι γαλοπούλες υπέρ των Χριστουγέννων. Σιγά μη συμβεί ποτέ αυτό το τραπεζικό σύστημα ε, παίρνει την έγκριση από τα κράτη-μέλη γιατί έτσι μόνο μπορούν ε, να λειτουργούν στην επικράτεια των κρατών μελών και στην ενιαία αγορά έχουμε ενιαίους κανόνες, έτσι. Αλλά για αυτό το θέμα δεν υπάρχει ε, αρμοδιότητα για να έχουμε ενίως ομοιόμορφους κανόνες για, το, για τη φορολογία γενικότερα δεν χρειαζόμαστε συνένεση, χρειαζόμαστε έναν ηγετικό ρόλο. Αν υπάρχει αποφασιστικότητα, αν υπάρχει ε, ε, ηγετικός ρόλος, ε, όπως είπα για τον πρόεδρο Μπαρόζο και άμα μου το ζητήσει θα το ξαναπώ, ε, όπως είπε λοιπόν στις 15 Δεκεμβρίου, αν δεν μας πάρουν ποτέ στα σοβαρά αν δεν έχουμε ηγετικό ρόλο και τι θα είναι η συνένεση, ο ελάχιστος κοινό παρανομαστής και ποιο είναι αυτό, Θέλουμε να δώσουμε όσο το δυνατόν γίνεται λιγότερα πράγματα Γιατί το φόρο των συναλλαγών ε, σε αντιπαραβολή με το τέλος σταθερότητας ε, ε, έχει μεγάλη παρουσιάζει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, επιπίας Βάσει όσα θα υπολογίσουμε το τέλος και επιπίεσε το, το φόρο. Δηλαδή, ε, εάν έχετε πολλές συναλλαγές θα έχετε και πολύ ψηλό φόρο και το αντίστροφο. Οπότε, Μην ξέρετε τι θα κάνουν οι ισχυρέ αγορέ. Ε, χρησιμοποιείτε το χρήμα για να έρθουν σε αντιπαράθεση οι κυβερνήσει. Ε, και αυτό ισχύει και στον τομέα των αγαθών και των υπηρεσιών. Ο κύριος Κασμάρικο Φίλιπ ήταν μαζί μου. Το είδαμε. Στην Μποτσουάνα. Μπράβο. Όλο Μπουρούντι μου έρχεται όταν σκέφτομαι την Μποτσουάνα. Επειδή είμαι και ομοφιλόφιλος ε, δεν, πρέπει να πάω εκεί πέρα γιατί θα με κλείσουν φυλακή. Αλλά τέλος πάντων, στην Μποτσουάνα ε, ε, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα μεσαίου εισοδήματο χώρα ε, που έχει τέτοιε συναλλαγέ. Ε, Διαμάντια έχει, νικέλιο έχει, χαλκό έχει, μα τα στέλνει όλα. Θα θέλαν αυτό το φόρο των συναλλαγών γιατί θα τους επιστραφεί ο φόρος. Χρειαζόμαστε ηγέτε. Ας του θυμίσουμε του Πρόεδρου Μπαρόζο τι είπε, α θυμίσουμε στου ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση τι είπαν. Όταν ήταν δημοφιλέ να κάνουν τέτοιε δηλώσει, τι κάναν και τώρα βλέπουν την αντίσταση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τι τράπεζε και υπαναχωρούν. Να του τα θυμίσουμε αυτά που είπαν ότι το ζητούν οι πολίτες και οι πολίτες έχουν ένα ισχυρότατο εργαλείο στα χέρια τους. Μην ξεχνάτε και τις εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με την ψήφο τους μπορούν να κάνουν την αλλαγή. Ε, είναι υπέρ αυτή τη θέση η κοινή γνώμη. Γι' αυτό δεν θέλουμε να χάσουμε εδώ το, το παράθυρο ευκαιρία. Μα δεν θα κλείσει. Είναι καταπληκτικό παράθυρο για την Ισπανική Προεδρία. Λοιπόν, αν χρειαστεί περισσότερο χρόνο, α πιάσει και την επόμενη Προεδρία. Το σημαντικό είναι να έχουμε τα αποτελέσματα αντί να συμβιβαστούμε με τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή και θα σκάσω τώρα. So, thank you very much. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κάσμαν. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά σας. Θυμίζω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 29 Απριλίου, μέρα 5η, στις 2 το απόγευμα. Και θα ψηφίσουμε στις 10 Μαΐου. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, σας προτείνω να κάνουμε τρία λεπτά διάλειμμα. Ε, μέχρι να έρθει κάποιος συνάδελφος που περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. dear colleagues, maybe we can... Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε. Θέλετε να περάσουμε και στο επόμενο θέμα στην μέση διαταξή. So, taking that we have... Έχουμε μόλις τρία τέταρτα για το επόμενο θέμα, πολύ σημαντικό και αυτό. Και σας προτείνω να συνεχίσουμε περιμένοντας τον κύριο Μπρόκ. Ερχόμαστε σε ένα σημαντικό θέμα τώρα ε, για το Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή μας. όπω γνωρίζετε, οι διαπραγματεύσεις για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης λαμβάνουν ε, χώρα μεταξύ των θεσμικών οργάνων αλλά και στο εσωτερικό των οργάνων. Στις 25 Μαρτίου, η κυρία Άστον κατέθεσε πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου που να ορίζει τη οργάνωση και λειτουργία της ευρωπαϊκής εξωτερικής δράσης. Για να ιδρυθεί αυτή η υπηρεσία χρειάζεται ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου που θα πρέπει να γίνει μετά από συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διαβούλευση με ε, το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή Εξωτερικών μαζί ε, με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ε, το συζητάει και με χαρά θα δεχτώ όταν φτάσει τον κύριο Έλμαρ Μπρόκ, τον εισηγητή, για την ανταλλαγή απόψεων εισηγητή της Επιτροπής Εξωτερικών. Θέλω να καλωσορίσω και τον κύριο Φερχόφστατ που συνεργάζεται ε, και αυτός με τον κύριο Μπρόκ. Είναι εδώ ο κύριος Φερχόφστατ. Αν θέλετε ελάτε στο Προεδρείο. And also I would like to η δική μας Επιτροπή θα γνωμοδοτήσει επίσης την έκθεση του κυρίου Μπρόκ για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και εμείς έχουμε ορίσει γιατί το συνάδελφο Φιλίπ Μα, ε, Κάσμαρεκ, συντάκτη γνωμοδότηση καλύτερα. Η έκθεση του κυρίου Μπρόκ θα βασίζεται σε ένα έγγραφο εργασίας και η συντάξη γνωμοδότηση είναι ο κύριος Φερχόφστατ Το έγγραφο εργασία έχει κυκλοφορήσει σε όλες τις ε, αρμόδιες επιτροπές. Έχει γίνει μεγάλη διαβούλευση στις 7 ε, Απριλίου ο κύριος Μπρόκ ήρθε στη συνεδρία των συντονιστών μας για να μας εξηγήσει το έγγραφο εργασίας και να ακούσει τις δικές μας ανησυχίες και μελήματα. Στο τέλος αυτής της συνεδρίασης συμφωνήθηκε η Επιτροπή να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για το έγγραφο εργασίας. Με χαρά Λέγω ότι πολλά από αυτά που προτείναμε συμπεριλαμβάνονται στην τελική εκδοχή των κειμένων, ωστόσο υπάρχει ένα βασικό στοιχείο που αφορά το στρατηγικό προγραμματισμό, ε, στο οποίο διαφέρουμε από ό,τι φαίνεται ακόμα. Προτείνω να αρχίσει η ανταλλαγή απόψε και θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Κάσ Μάρεκ, συντάκτη γνωμοδότησή μας. Παρακαλώ, έχετε μέσα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα γιατί έχει αλλάξει λίγο ο τρόπος εργασίας μας ε, από την κλασική λειτουργία της Επιτροπής Ανάπτυξης και μετά. Θέλω να ευχαριστώ ε, στις όλους εκείνους που συμμετείχαν σε αυτή την υπόθεση, την κυρία Εύα Ζολή, που εκπροσώπησε την Επιτροπή ε, μαζί μου ε, κατά τη διάρκεια των επαφών που είχαμε. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συντονιστές που αφιέρωσαν ξεχωριστή συνεδρίαση αποκλειστικά σε αυτό το θέμα αλλά και τη γραμματεία που εργάστηκε ε, στενά για το θέμα αυτό. Κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή μας για την Εξωτερική Δράση Επικεντρώθηκε βέβαια στα θέματα που άπτονται της ανάπτυξης. Ε, μας, ε, δεν μας ενδιαφέρει το σύνολο ε, της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Έχουμε τη σκοπιά της ανάπτυξης που μας απασχολεί περισσότερο. Και εκεί βλέπω διάφορα στοιχεία. Σήμερα θα πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση, Κιζόλη. και στο βαθμό του δυνατού θα προσπαθήσουμε να το ε, γράψουμε και στο κείμενο. Δεύτερη σημαντική διάσταση είναι η επίδραση των επιτρόπων ε, στον προγραμματισμό και την εφαρμογή όλων αυτών για να αποφύγουμε ενδεχόμενες αντιφάσεις μεταξύ των πολιτικών στόχων και των ε, στόχων ε, όπου δαπανούμε χρήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι ε, θα πρέπει οι επίτροποι να έχουν πρόσβαση στα μέσα αυτά, να μπορούν να επηρεάζουν τις υπηρεσίες δηλαδή που θα εργάζονται για την εξωτερική δράση. Οι επίτροποι δεν μπορούν να στερούνται αυτού του δικαιώματος πραγματικών εργαλείων μέσων εργασίας και μια τέταρτη διάσταση ε, παραμένουν εκεί οι διαφορές, δεν είναι πολύ μεγάλες. Αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έχουμε συντρέχουσες αρμοδιότητες. Και μπορούμε να έχουμε και κάποιες διαφορές απόψεων, δεν συμφωνούμε πάντα με την ε, κατεύθυνση και την έμπνευση που δίνεται ε, σε αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι συνομιλητής για μας και θα πρέπει να πάρει την απόφαση ως συλλογικό σώμα. Αυτή θα είναι η τελική απόφαση. Όπως είπε η Πρόεδρος, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που εκκρεμεί και δεν έχει λυθεί ακόμα και αυτό είναι ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός ή η ερμηνεία του ε, ο καθορισμός ε, των αναπτυξιακών μέσων, πώς θα γίνουν όλα αυτά και πώς θα μπορέσουν οι επίτροποι να χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα. Ε, κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι ακριβώς να φτάσουμε σε κοινή θέση, διότι το Κοινοβούλιο κανονικά θα πρέπει να διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο και χρειάζεται ενιαία θέση είναι πολύ σημαντική αυτή για να έχουμε διαπραγματευτική ισχύ και ατού στα χέρια μας. Αυτά και προσβλέπουμε σε αυτή τη συνεργασία. Ξέρω ότι και οι συντονιστές επιθυμούν και οι συντάκτες και οι συγητές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει στα πολωνικά η Πρόεδρος. Περιμένοντας τον κύριο Μπροκ, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκίφερ Χόφστατ να μας εξηγήσει τις απόψεις του για την ίδρυση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Στα γαλλικά, ο κύριος Φερχόφστατ, ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία συντάξει Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων να συμμετέχω σε αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής σας, ίσως θα πρέπει να γνωρίζουμε το εξής και να υπογραμμίσουμε πρώτα απ' όλα ότι ο κύριος Μπροκ και εγώ αποφασίσαμε να κάνουμε μία έκθεση με κοινέ τροπολογίες. Δηλαδή θα είναι ακριβώς οι ίδιες τροπολογίες που θα κατατεθούν ε, στην Επιτροπή Εξωτερικών και στην Επιτροπή ε, Συνταγματικών Υποθέσεων Πράγμα που ενισχύει νομίζω ότι θέση ε, τη διαπραγματευτική του Κοινοβουλίου στη διαπραγμάτευση με τις άλλες, ε, τα άλλα θεσμικά όργανα, την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ένα αυτό. Δεύτερον, αφετηρία του κυρίου Μπροκ και μου ε, όταν ε, κάναμε την έκθεση. Το τελικό κείμενο που έχετε στις 20 Απριλίου έχει ημερομηνία. προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη όσο γίνεται περισσότερο τις δικές σας ε, προτάσεις και τα σχόλια. Στην αρχή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θελήσαμε να είναι φιλόδοξη, να μην περιορίζεται δηλαδή σε μια διπλωματική υπηρεσία, να είναι σολάν ας πούμε, ε, πάνω από χίλιοι διπλωμάτες που κάνουν αυτό που έκαναν και στο παρελθόν. Δεν λέει αυτό η συνθήκη. Στο άρθρο 21 ορίζει ξεκάθαρα ότι θα πρέπει όλες οι πολιτικές εξωτερικής δράσης να ενταχθούν σε αυτή την υπηρεσία. Να συνενωθούν και να μην είναι ένα διπλωματικό σώμα βελτιωμένο τρόπο την αυτή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Και γνωρίζετε ότι το άρθρο 27 της συνθήκης, 21 διορθώνει ο κ. Φερχόφστατ, στη σελίδα 3, ε, απαριθμεί ε, όλες τις αποστολές και τα καθήκοντα τα οποία θα πρέπει να επομίζεται ε, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης και βέβαια εκεί είναι και η αναπτυξιακή συνεργασία. Αυτή είναι λοιπόν η αφετηρία μας. Να έχουμε μια υπηρεσία εξωτερικής δράσης πιο φιλόδοξη και όσο γίνεται πιο συνεκτική. στη συνέχεια, ένα τρίτο στοιχείο μετά από την αφετηρία και το, σημείο κίνησης και εμείς το 90% των μέσων και το 90% των πόρων προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ουσιαστικά είναι τμήμα, ε, μονάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Γιατί είναι στο τμήμα 3 του Γενικού Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως γνωρίζετε το τμήμα 3 είναι ε, εκείνο που αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για ποιο λόγο. Διότι το τμήμα 3, ε, η κατηγορία 3, είναι πραγματικά στην καρδιά της κοινοτικής δράσης και πολιτικής. Συμπεραβάνει όλες τις δράσεις της Ένωσης, στη λεγόμενη κατηγορία 1, 2, 3, 4 κτλ. Ε, και εκεί ακριβώς ε, την εξωτερική πολιτική Και το ε, επόμενο που μας απασχόλησε είναι να έχουμε ε, μια φιλόδοξη υπηρεσία εξωτερικής δράσης και αυτή να τη συνδέσουμε, επαναλαμβάνω, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα ε, έτσι θα είμαστε και πιο συνεκτικοί και πιο συνεπείς. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο αυτή υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο εσωτερικό της εξωτερικής δράσης να συνδεθεί και η Επίτροπος που είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, η Επίτροπος Γειτονίας, Επίτροπος ε, ε, ε, Ανθρωπιστικής Βοήθειας και η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος. Τα προβλήματα αρχίζουν τη στιγμή που θέλει κάποιος να κάνει μια φιλόδοξη υπηρεσία εξωτερικής δράσης εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα, προφανώς. Και πρώτη φορά θα γίνει κάτι τέτοιο. Για πρώτη φορά θα δημιουργηθεί μια υπηρεσία σημαντική όπως είναι αυτή, εκτός της μεθόδου ε, της κοινοτικής και της κατηγορίας 3, γιατί είναι η μετάφραση της κοινοτικής μεθόδου στον προϋπολογισμό. Ε, le, le, le ποια είναι η κατάσταση τώρα, τη γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Ε, εγώ είμαι νεόφυτος ε, σε αυτά τα θέματα. Ε, πώς έχει η κατάσταση για τη συνεργασία μέχρι τούδε. Μέχρι τούδε. Ε, όλα τα αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ανάπτυξη που κάνει τον προγραμματισμό και στη συνέχεια η Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων ασχολείται με την υλοποίηση ε, υπό την αιγίδα ενός επιτρόπου. Βέβαια υπήρξαν και δυσκολίες, έτσι, ορισμένες φορές. Εγώ είχα το μεγάλο πλεονέκτημα να είμαι στενός φίλος και πολιτικός φίλος του ε, Λουί Μισελ, του προηγούμενου επιτρόπου ε, για τα αναπτυξιακά θέματα και μου διηγήθηκε πολλές συγκεκριμένε υποθέσεις όπου παρότι στον προγραμματισμό είχαμε αποφασίσει να κάνουμε κάτι, επί του τόπου κάναμε κάτι εντελώς διαφορετικό ή τίποτα. Ε, λέγαμε ναι εντάξει ωραίος ο προγραμματισμός εγώ είμαι αξιωματούχο επιτροπής που πρέπει να αποφασίσει για τι δαπάνε, αλλά δεν κάνω τίποτα γιατί δεν έχω λεφτά ή γιατί έχω άλλε προτεραιότητε. Με τωρινή κατάσταση δεν είναι προφανέ έτσι να ε, ε, είναι συνεκτική η γιατι εχω αλλε προτεραιοτητες με τωρινη κατασταση δεν ειναι προφανε ετσι να ειναι συνεκτικη η πολιτικη για τη συνεργασία. Αυτά συμβαίνουν γιατί στον προγραμματισμό τη ΓΑΜΑ ε, και στον προγραμματισμό της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων ε, τι συμβαίνει. Έχουμε δύο συναρμόδιε υπηρεσίες που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την αιγίδα του αρμοδίου επιτρόπου, δηλαδή του Επιτρόπου για τα αναπτυξιακά ζητήματα. Για τον προγραμματισμό, το ξέρετε, ότι τα δύο πρώτα στάδια γίνονται από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ανάπτυξης ε, και ε, το τελευταίο από την EuroPaid. Έτσι έχει κατάσταση τώρα. Τι γίνεται τώρα με την πρόταση της κυρίας Άστον. Περιπλέκεται έτσι περαιτέρω το θέμα. Ε, αφενός φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυρία Άστον συμπόγραψαν συμφωνία που περιπλέκει την κατάσταση. Γιατί? Ε, γιατί τώρα θα έχουμε τρία διαφορετικά στάδια προγραμματισμού. Πρώτον, θεματικός προγραμματισμός ε, από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ε, ανάπτυξης. Μετά, προγραμματισμός γεωγραφικού χαρακτήρα από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και μετά θα επανέλθει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση από τη ΓΔ EuroPaid. Περιπλέκεται λοιπόν η υπόθεση ήδη υπάρχουν αντιφάσει όπως έχει τώρα η κατάσταση, θα οξυνθούν περαιτέρω ε, με τα ε, ε, τους νέους κανόνες. Εδώ και 48 ώρες παίρνω επιστολές, email και όχι μόνο εγώ και εσείς. Σωρία λοιπόν επιστολών για να εξηγήσουν την πρόταση που έκανε η κυρία Άστον σε συνεργασία με την Επιτροπή Χτες το βράδυ εγκρίθηκε η πρόταση από το Συμβούλιο και εξηγείται ε, πού ελοχεύει ο κίνδυνος, ε, πού ε, ενδέχεται να δυσλειτουργεί στο σύστημα ή εν πάση περιπτώσει να έχουμε οξυμένες αντιθέσεις σε σχέση με το παρελθόν. Ε, ποια είναι η πρότασή μας λοιπόν λόγω του ότι ε, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ανήκει στο τμήμα 3 και άρα είναι συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χοντρικά ισχύουν τα ίδια με σήμερα. Ε, δηλαδή, η γάμα δέλτα ε, ανάπτυξης ε, μπαίνει στα χωράφια της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, η οποία όμως συνδέεται με την Επιτροπή και ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και άρα για τη διαχείριση και το συντονισμό, ο αρμόδιος για την ανάπτυξη επίτροπος ανήκει σε αυτή την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Δεύτερον, ε, για την εκτέλεση αρμόδια είναι η Europaid. Και η Επιτροπή, είναι και η Europaid, έτσι, αλλά άλλο τμήμα της Επιτροπής που ασχολείται με την υλοποίηση. Οπότε, η κατάσταση που ε, προκύπτει από την πρόταση μας, επανέρχεται στην ε, τωρινή κατάσταση. Εφόσον, ξαναλέω, η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η εκτέλεση, η υλοποίηση γίνεται από την Europaid. Άλλο κομμάτι τη Επιτροπή. Αυτό ήταν το πρώτο σημείο. Δεύτερον, οι δύο υπηρεσίε ε, υπάγονται στην αρμοδιότητα του ιδίου επιτρόπου. Τι σημαίνει αυτό. Στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, όλοι όσοι ασχολούνται και με τα οριζόντια θέματα και με τα γεωγραφικά έτσι, σε εισαγωγικά θέματα ε, τα, που σχετίζονται με την ανάπτυξη όλοι υπάγονται στον Επίτροπο. Και ε, η εκτελεστική αρχή όμως η Europaid τελεί υπό την αιγίδα του ίδιου Επιτρόπου. Ε, ρίστο εμπαροδότη, μες στην πρόταση της κυρίας Άστον τα οριζόντια και τα γεωγραφικά εισαγωγικά θέματα. Λυπάμαι, αλλά ε, έχουν ένα δυσδιάκριτο όριο. Μα το, το ίδιο πράγμα είναι. Στην ίδια πρόκληση καλούμεθα να ανταπεξέλθουμε. Είναι λίγο τεχνητή η διάκριση, δηλαδή να μην ανήκουν στην ίδια γενική διεύθυνση, όπως αντίθετα, ε, ε, όπως προτείνει μάλλον η κυρία Άστον. Ε, και το ίδιο για τα τρία αυτά στάδια. Ε, στάδιο 1, 2, 3, ο προγραμματισμός δηλαδή. Γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση για την Ανάπτυξη της Εξωτερικής Δράσης και θα υλοποιηθούν από τη Europay τα στάδια 4 και 5 δηλαδή, αλλά η Europay στην Επιτροπή ανήκει επίσης. αν εκτελεστεί 100% η πρόταση που εμείς υποβάλαμε, εγώ πιστεύω ότι το ισχύον σύστημα θα εξακολουθήσει να ισχύει. Με τη μόνη διαφορά ότι η γάμα δελτα θα ανήκει στην υπηρεσία εξωτερική δράση που ξαναλέω συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο αρμόδιο για την ανάπτυξη ε, επίτροπο ε, και αυτό που ασχολείται με την γειτονία και την ανθρωπιστική βοήθεια θα ε, συνεργαστούν με την κυρία Άστον. Και οι λοιποί συγκητές πιστεύω έχουν παρόμοιες απόψεις δεν μπορούμε τώρα να συνδέσουμε εδώ την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τουλάχιστον από δημοσιονομικής απόψεως. Οπότε οτιδήποτε σχετίζεται με την ανάπτυξη νομίζω πρέπει να είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρχει καλός συντονισμός. Δεν ε, υποστηρίζω την πρόταση της ε, στον αλλού τα οριζόντια ε, θέματα, αλλού τα γεωγραφικά ζητήματα το σημαντικό είναι να είναι συνεκτική η αναπτυξιακή μας πολιτική. Αυτό έχει ε, θεμελιώδη σημασία για να είναι και αποτελεσματικές οι δράσεις μας και για να ε, κατοχυρώσουμε ότι οι προσπάθειες που καταβάλουμε και τα κονδύλια που διαθέτουμε θα έχουν αυτά αποτελέσματα. Κάτα τα λοιπά. Στην ε, τελευταία εκδοχή με ημερομηνία 20 Απριλίου. Ε, νομίζω συμπεριλαμβάνονται όλες ε, οι παρατηρήσεις που διαβίβασε στον κύριο Μπρό και στον υποφαινόμενο η Επιτροπή σας. Αλλά και πάλι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι συνάρτηση της ε, βούλησης του Συμβουλίου και της Επιτροπής, αλλά κυρίως του Συμβουλίου, να συμφωνήσει με εμά για τα θέματα αρχή, Δηλαδή, χοντρικά, ε, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, ανήκει, υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θα είναι στο τμήμα 3 ή όχι. Αν ναι, νομίζω ότι είναι καλή η εισήγησή μας για να είναι συνεκτική αναπτυξιακή πολιτική. Εάν είναι αρνητική όμως η απάντηση σε αυτό το ερώτημα και πάλι εγώ ε, θα ταχθώ υπέρ ε, του να αναλάβει εκ νέου η Επιτροπή όλες τις αρμοδιότητες και θα αφήσουμε με περιορισμένο πεδίο δράση στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και δεν μπορούμε να τα έχουμε και τα δύο. Δηλαδή ισχυρή φιλόδοξη υπηρεσία εξωτερικής δράσης που θα τα αναλάβει όλα και ταυτόχρονα να την αποσπάσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν γίνεται αυτό, καταπατούμε την ενωσιακή μέθοδο έτσι. Ίσως υπερβάλλω έτσι συνήθως. Τέλος πάντων, είναι ένα μικρό ε, δημοσιονομικό πραξικόπημα, έτσι, αν ε, το κάνουμε αυτό και πρέπει να αποφύγουμε την παραβίαση της ενωσιακής μεθόδου. Ευχαριστώ. Μετά τα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν πριν να αρχίσει η συζήτηση με τους ε, βουλευτές. Χρήσιμο θα ήταν λοιπόν να ακούσουμε τη θέση και στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς εξηγεί τη διαφορά μεταξύ της πρότασης Άστον και της πρότασης Φερχόφστατ κάθετος Μπροκ. Η Κομισιόν, λοιπόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες. Πολλά από τα σημεία τα οποία τέθηκαν έχουν ήδη ακουστεί ξανά και ξανά σε πολλές συζητήσεις. Θέλω απλώς να εστιάσω στα τέσσερα σημεία που αναφέρθηκαν στην αρχή και σε ένα-δύο έξτρα σημεία που είπε ο κ. Φερχόφστατ. Για τα τέσσερα σημεία. Η στρατηγική προτεραιότητα για την πολιτική σημασία της ανάπτυξης. Όχι μόνο συμφωνούμε, αλλά όλη η προσπάθεια έχει νόημα για να αναβαθμίσουμε την αναπτυξιακή πολιτική. Από αυτό που σήμερα είναι απλή διανομή χρήματος ε, σε κάτι πολύ πιο στρατηγικό. Επομένως, η αναπτυξιακή πολιτική θεωρείται ε, σημαντικό τμήμα της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος αυτού. Δεύτερον, για την ε, επιρροή της ε, Επιτροπής και για να αποφύγουμε τις αντιφάσεις. Σήμερα η κατάσταση είναι κατακαιρματισμένη και εξαρτάται πολύ από τα διάφορα μέσα και εργαλεία και λιγότερο από τις πολιτικές. Η πρόταση λοιπόν μιλάει για το γεγονός ότι ο Επίτροπος Ανάπτυξης είναι υπεύθυνο και καθορίζει από την αρχή το περιεχόμενο των πολιτικών. Τώρα για την πρόσβαση στο μέσο. Για πρώτη φορά εδώ και δέκα χρόνια, τα δύο βασικά μέσα, τα δύο βασικά εργαλεία, δηλαδή όλοι οι γεωγραφικοί τομείς ε, για την ανάπτυξη καλύπτονται για, την προγραμματική περίοδο, για τον προγραμματισμό μάλλον από ένα και μόνο επίτροπο. Ένας και μόνο επίτροπος είναι αρμόδιος. Όχι δύο-τρεις επίτροποι. Αυτό μας το ζητήσανε και πολύ σωστά μας το ζήτησε και το Κοινοβούλιο. Και τώρα έχουμε τον ίδιο επίτροπο που είναι υπεύθυνο και για το EDF και για το DCI, το Μέσο για την Αναπτυξιακή Συνεργασία. Τώρα, η διαδικασία λήψη των αποφάσεων. Η Κομισιόν και το Σώμα των Επιτρόπων, λέμε, πρέπει να αποφασίζει. Αυτό λέει η πρόταση, ότι για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν ε, στα πλαίσια του DCI και EDF και το μέσου γειτονίας, γειτονίας παρουσιάζονται στο Σώμα των Επιτρόπων αυτές οι αποφάσεις από την α, Αντιπρόεδρο κάθετο είπα το εκπρόσωπο. Επομένως, τα τέσσερα σημεία λαμβάνονται υπόψη από την πρότασή μας και συμφωνούμε απόλυτα. Υπάρχουν τώρα ένα-δύο σημεία που έθεσε ο κύριος Φερχόφσταντ. Ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα όπως έχει η κατάσταση. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει κατακαιρματισμός μέσων και εργαλείων, ότι εξαρτώμαστε από τα μέσα και από τα εργαλεία και όχι από τις πολιτικές. Αυτό είναι καθημερινό ψωμοτήρι για μένα. Ε, στην αναπτυξιακή πολιτική. Ε, για να γίνει, τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να την κάνουμε πραγματικά καθολική και παγκόσμια. Ε, γιατί σήμερα με τα εργαλεία και τα μέσα περιθωριοποιείται. Και σήμερα είναι η ευκαιρία για να καταστήσουμε αυτή την πολιτική τμήμα της απάντησης στην κρίση Αναβαθμίζουμε έτσι όλες τις, αναβαθμίζουμε την αναπτυξιακή πολιτική. Νομίζω ότι με αυτή την κατάσταση. Και δεν διαιωνίζουμε τη σημερινή κατάσταση. Έπειτα, ο προγραμματισμός με τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα, με τα στρατηγικά προγράμματα τα κτλ. Αυτά μπορούν να συνεισφέρουν ε, σε ένα μείγμα πολιτικών ε, και σε ένα μείγμα εργαλείων από την αρχή για να εφαρμοστούν αυτά τα μέσα ε, και γίνονται καλύτερο εργαλείο για την, για το, στα χέρια του Επιτρόπου Ανάπτυξης. Θέλουμε να κάνουμε διάκριση τώρα μεταξύ των, προγραμμάτων, ε, των εργαλείων συγγνώμη, προγραμματισμού και μη προγραμματισμού. Τα εργαλεία προγραμματισμού είναι τα γεωγραφικά. Στην αρχή του κύκλου αποφασίζουμε για τα ποσά. Αυτό είναι προνόμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με, το, με τη χώρα αποφασίζουμε πού εστιάζουμε τις προσπάθειές μας. Ε, έχουμε κοινή στρατηγική. Μέχρι στιγμής τα έγγραφα στρατηγικής αναχώρα ήταν έγγραφα για να κινητοποιήσουμε τον κόσμο για να ξοδέψει τα χρήματα και όχι για να καταστήσει, να δημιουργήσει στρατηγική. Και δεύτερον, ε, έχουμε τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα, πώς θα ξοδευούν τα ε, χρήματα ανά περίοδο. Τα θεματικά προγράμματα κάνουν όμως κάτι διαφορετικό. Δεν, δεν έχει να κάνει με τη χώρα και τον προγραμματισμό, αλλά ε, με την υποστήριξη δραστηριοτήτων, ε, επένδυση στις, ε, στην υγεία, στους ανθρώπινους πόρους κτλ. Δεν προσθέτουμε χρήματα στις χώρες, αλλά θέλουμε σε παγκόσμιο επίπεδο να προωθήσουμε πρωτοβουλίες, συγχρηματοδότηση δράσεων, ας πούμε, ε, με τις οργανώσεις του ΟΗΕ, έρευνα στην γεωργία κτλ. κτλ. Αυτό δεν επηρεάζεται καθόλου. Αντίθετα, νομίζω ότι αυτά είναι τα ιδανικά εργαλεία και το ξέρει πολύ καλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί το Κοινοβούλιο ε, βρίσκεται στην ρίζα αυτών των προγραμμάτων, ε, συμπληρώνουν λοιπόν ε, τις πολιτικές. Τώρα, έχουμε την εφαρμογή των πολιτικών κάτι που είναι τελείως ξεχωριστό. Επομένως δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σταματώ εδώ γιατί όλα τα υπόλοιπα ε, είναι τμήμα ε, μιας συζήτησης που έχει γίνει πολλές φορές και σε διάφορα φόρουμ. Ε, χθες ε, το Συμβούλιο έφτασε σε πολιτική συμφωνία για διάφορα θέματα. Κάποια από αυτά σας ενδιαφέρουν, κάποια όχι. Μπορώ να σας πω πάντως ότι σας ενδιαφέρει. Σταματώ εδώ λοιπόν ε, και είμαι έτοιμο να απαντήσω οποιασδήποτε ερωτήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπροκ που μας διαθέτει το χρόνο του για να έρθει στην Επιτροπή. Να του δώσω το λόγο. Ε, ίσως θέλει να προσθέσει δύο λόγια και συνεχεία αρχίζει η συζήτηση. Και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, το πρώτο το αγκλαστικό είναι πάντα να στρέφομαι προς τα δεξιά. Τι να κάνω κι εγώ. Ε, τώρα δεν θέλω να σας κάνω ε, μεγάλη τοποθέτηση, γιατί δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Φερχόφστατ. συγγνώμη για την καθυστέρηση, με καθυστέρηση η Επιτροπή Εξωτερικών. Δεν θέλω επικαλύψεις να συζητήσουμε. Αν θέλετε να σας ενημερώσω για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα το απόγευμα με το Συμβούλιο τους ε, υπαλλήλους κυρία Άστον και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συζητήσαμε και θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτικό έλεγχο, όχι μόνο τα δημοσιονομικά δικαιώματα, ε, αλλά βεβαίως δεν υπάρχουν πλέον άλλες δυνατότητες. Πρέπει να κινηθεί έτσι το Συμβούλιο. Κυρία Άστον. Ε, είπε κάποια πράγματα, αλλά στα πολιτικά ε, ζητήματα και στον πολιτικό έλεγχο και στον διοικητικό έλεγχο έχουμε περιθώριο χειρισμών και έχουμε και ένα μνημόνιο συνεννόηση που μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς ε, αποφασίζονται κάποιες στρατηγικές όταν ε, κάποιες εντολές και να υπάρχει προηγούμενη διαβούλευση με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές που είναι αρμόδιες και για τον πρακτικό έλεγχο είναι αυτό σημαντικό και ό,τι έχει να κάνει με τα έγγραφα στρατηγικής, με συνθήκες και συμβάσεις, με ε, εντολές, με διαχείριση κρίσεων, με αποστολές και ε, λήψη αποφάσεων με στο αρμόδιο όργανο και σε διαβούλευση προηγούμενη επαναλαμβάνω με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Όλα αυτά είναι θέματα πολύ σημαντικά και στην πράξη ε, αφορούν και την αναπτυξιακή συνεργασία και την ε, εξωτερική πολιτική. Αν δεν το είπε αυτό ο Γκί θα ήθελα να το συμπληρώσω αυτό, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό. Και σε θέματα, ε, να βρούμε μια κρίσιμη μάζα για να ε, μπορούμε να διαμορφώσουμε πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Α, συγγνώμη. Γιατί ήρθα εγώ στην Επιτροπή Ανάπτυξη από την Επιτροπή Εξωτερικών, γιατί καμιά φορά σου δίνει και κανένα κομμάτι σοκολάτα εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Thanks to the Αυτά είναι τις γραμματείας θέματα. Α, βρήκαμε το μυστικό να σε κρατήσουμε τρεις ώρες εδώ πέρα χωρίς να διαμαρτύρεσαι. Υπάρχουν ερωτήσεις, σχόλια. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μαντεβίση, κύριε Φερχώστατ, κύριε Μπρόκ. Ευχαριστώ και δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι ειδικό. Αλλά όσα περισσότερα ακούω, τόσο πιο πλεγμένα μου φαίνονται όλα αυτά. Να σας πω πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ. Στην Επιτροπή Ντεβε και στις ΜΚΟ που ασχολούνται με τα αναπτυξιακά θέματα υπάρχει αντίληψη ότι θα υποβαθμιστεί ο ρόλος της αναπτυξιακής πολιτικής ε, και η εξάλληψη της ε, φτώχειας, ε, οι προσπάθειες που γίνονται για την εξάλληψη της φτώχειας θα μειωθούν και θα χρησιμοποιηθεί η αναπτυξιακή βοήθεια μόνο, μόνο μέσω της εξωτερικής πολιτικής. Σοβαρές ανησυχίες δηλαδή. Επίσης, χτες ο κύριος Μανσεβίση, δεν ξέρω ή εσείς έχετε δει το σχετικό δημοσίευμα, τη, συγγνώμη, τη σχετική νομική γνωμοδότηση που κυκλοφόρησε χθες, ε, όπου αμφισβητείται η πρόταση της Βαρόνης Άστον σε σχέση με την συνθήκη. Αν θέλετε να σας το διαβάσω κιόλας. Uh, Λέει λοιπόν για την υπηρεσία εξωτερική δράση που άνευ αποκτά έλεγχο για την, ε, την αναπτυξιακή πολιτική και τον σχετικό προπολογισμό ότι υπάρχει ένα μείγμα κυβερνητικών ε, και ενωσιακών πολιτικών και είπαμε ότι χρησιμοποιείται για λόγους εξωτερικής, για σκοπιμότητες εξωτερικής πολιτικής πλέον η πολιτική ε, για την αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, από αυτά που είπε ο κ. Μαντσεβίση καταλαβαίνω ότι ο Επίτροπος Αρμόδιος για την Ανάπτυξη πρέπει να εμπλακεί στον ε, άμεσο έλεγχο και καθοδήγηση και στα πέντε στάδια του προγραμματισμού ε, να έχει ένα ισχυρό ρόλο χωρίς επικαλύψεις μέσα στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης έτσι η ανάπτυξη θα μεταβιβαστεί ε, στις αρμοδιότητες, ε, θα υπαχθεί μάλλον ε, στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Όταν ε, αναθεωρηθεί η υπηρεσία εξωτερικής δράσης που προτείνεται για το 2012 λέει εδώ ότι πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε θα αναθεωρηθεί και ο προγραμματισμός ε, και όχι μόνο από την οπτική γωνία της εξωτερικής πολιτικής αλλά λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Επίσης, χρειαζόμαστε ένα εχέγγυο ούτως ώστε να ε, πληρωθούν φιλόδοξοι στόχοι και να τηρηθούν υποσχέσεις για την απτυξιακή πολιτική. Οι δεσμεύσει ε, άκρα παραδείγματο χάρη για την αποτελεσματικότητα τη ε, βοήθεια, η δήλωση του Παρισίου. αυτό νομίζω θα καλύψει ανησυχίε κάποιων μη κυβερνητικών οργανώσεων και βουλευτών. Το τελευταίο σας το σχέδιο, κύριοι Μπρόκ και Φερχόφστα, δεν το έχω δει. Αλλά αυτό που είδα και όπως το συζητήσαμε στην ε, πολιτική μου ομάδα ε, και ε, εδώ μιλώ και εξ ονόματος της ομάδας μου, SND, υπήρχε αναφορά σε σε προσωπικότητε που θα έχουν σχεδόν πολιτικό χαρακτήρα και θα επικουρούν την αντιπρόεδρο καθώς ε, είπα του εκπρόσωπος ε, την κυρία Άστον δηλαδή. Για να μην είμαι κοινικό, γιατί ποτέ δεν είμαι κοινικό, ε, νομίζω ότι οι αναπληρωτές, οι τέσσερις διευθυντέ αυτοί δεν θα αναλάβουν το ρόλο που νόμιζαν. Θα είναι εξαιρετική σύμβουλη της Ευαρώνης Άστον αυτή η σχεδόν ε, πολιτική συμβουλή ε, θα είναι η συνταγή για την αποτυχία. Ε, αν θέλετε τη δική μου γνώμη. Ούτε ο πρόεδρος Μπαρόζο δεν έχει τέτοιους σύμβουλους, έχει αντιπροέδρους ας ε, δώσουμε στην Αντιπρόεδρο και ύπατη εκπρόσωπο την εξουσία που χρειάζεται, ε, ας δώσουμε στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης τη δύναμη που χρειάζεται και δεν θα υποβαθμιστεί ο ιστορικός και σημαντικός ρόλος που παίζει ε, η βοήθεια στην αναπτυξιακή μας πολιτική. και δεν πρόκειται να υπαχθεί αναπτυξιακή πολιτική σκοπιμότητα εξωτερικής πολιτικής. Ευχαριστώ κύριε Κάσμαν. Um, thank Βέρμαν, um, είναι γεγονός ότι η Επίτροπος θα έχει και το DCI και το ETF, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και το Μέσο της Αναπτυξιακής ε, Βοήθειας. Είναι μεγάλη ε, επιστοδρόμηση και είναι λιγότερο αριστοκρατική ευγενής η πρόταση από την ίδια τη Βαρόνη, την Επίτροπο που είναι ευγενής πώς να το πω, δηλαδή δεν γίνεται λόγος πουθενά για ευθύνη. Πρόκειται για καθοδήγηση και για υποπτία, που είναι άλλο πράγμα στην πρόταση. Δεν βλέπω πουθενά την ευθύνη εγώ, την υπευθυνότητα τη επιτρόπου, της, ή του επιτρόπου του ίδιου. Εποπτεία και καθοδήγηση, χαιρετίσματα. Είναι αρκετό αυτό. Το πρόγραμμα ε, της, Άστον για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράσης ε, είναι πάρα πολύ συγκεχημένο. Και ποιο θα τα κάνει αυτά και ποιο θα τα χρηματοδοτεί επικρατεί σύγχυση στην όλη πρόταση μεταξύ ε, του κύρους της αρχής και της ευθύνης. Το κύρος της κυρίας ε, Άστον, τι σημαίνει ότι θα είναι υπό, υπευθύνη της και αυτό υπό την ευθύνη της κυρίας Άστον είναι λάθος έτσι όπως το προτείνεται. Και θα ήταν οπισθοδρόμηση κατά 50 έτη τουλάχιστον όταν η αναπτυξιακή πολιτική ήταν ένα εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Και σήμερα ασκείται πολύ μεγάλη κριτική κατά της αναπτυξιακής πολιτικής ότι δεν λειτουργεί, ότι τα πάντα έχουν αβαγίσει. Γιατί ένας από τους μεγαλύτερους λόγους είναι ότι ποτέ δεν ε, πήραν σοβαρά την αναπτυξιακή πολιτική και πολλοί δικτάτορες διατηρήθηκαν στα πράγματα και αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι το εμπόριο και λιγότερο οι νόμιμες ε, ε, προσδοκίες των λαών και για διάφορους λόγους αποφασίσαμε ότι εντάξει ε, ας ε, αρκεστούμε και σε λιγότερη αναπτυξιακή πολιτική. Δεν νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτή τη ε, κατάσταση που είναι πιο σημαντική οι από τη μείωση της φτώχειας. Όχι, δεν θα πρέπει να κυριαρχούν στην ανάπτυξη σκέψη εξωτερικής πολιτικής. Και είναι αντίφαση αυτό με τη συνθήκη την ίδια της Λισαβόνας Ε, και η ΣΥτσΕ και η Κόνκορτ ζήτησαν ε, και νομική γνωμοδότηση για να εντοπιστούν στην πρόταση της Άστον οι αντιφάσεις με τη συνθήκη. Για μένα ε, η ενοποίηση των υπηρεσιών δεν είναι από μόνο του επικίνδυνο. Δεν φοβάμαι καθόλου εάν η Επίτροπος στην εξωτερική δράση έχει την ίδια την ευθύνη της και για τον προγραμματισμό, όπως είπε ο Μάικλ σωστά, και για τις πέντε φάσεις της αναπτυξιακής πολιτικής, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να έχει αυτή την υπηρεσία ε, ενωμένη με την αναπτυξιακή βοήθεια. Αλλά αν είναι τα πράγματα τόσο σαφή και, σαφή και αόριστα και συγκεκριμένα, φοβούμε ότι δεν θα ε, δουλέψει, δεν θα λειτουργήσει σωστά και είναι συνταγή για συνέπεια στις πολιτικές και για σύγκρουση. Αυτό ακριβώ λοιπόν είναι η πρόταση ε, ε, ε, που θέλουν να αποφύγουν και να αλλάξουν ο, ο Φερχόφστατ και ο Μπροκ προς το καλύτερο και χαίρομαι πάρα πολύ που οι προτάσεις που κάνετε και μας παρουσιάζετε έχουν εξελιχθεί πολύ από τα πρώτα βήματα, τα αρχικά που είχατε κάνει. Μπορεί στην αρχή να είχαμε κάποιες μικροδιαφωνίες για ίσονο σημασία ζητήματα. Αυτό που εσείς προτείνετε είναι να υπάρχει επίτροπος αρμόδιος και η είπατε εκπρόσωπος να έχει το κύρος, ξέρω να έχει την πολιτική ε, ευθύνη, εν πάση περιπτώσει. Ναι, εντάξει. Και να έχει αρκετό κύρος για να μπορεί να λειτουργεί ως είπατε εκπρόσωπος. Για κάθε επίτροπο βέβαια αυτό και στο εσωτερικό της υπηρεσίας. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σαρχεντίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λέει η πρόταση της κυρίας Άστον ότι η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και οι υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα κάνουν αμοιβέ διαβουλεύσεις. Ένα λεπτάκι. Περιμένω κάποιος έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση εκεί στο Προεδρείο. Λέει λοιπόν ε, η πρόταση της κυρίας Άστον ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα διαβουλεύεται με τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκή Επιτροπής ε, και το αντίστροφο ε, στο υπέροχο κεφάλαιο που τυκλοφορείται συνεργασία άρθρο 3,2. Μ' αρέσει η λέξη συνεργασία και η λέξη διαβούλευση αλλά προτιμώ λέξεις όπω και τώρα απηχώ την παρέμβαση του συναδέλφου από το S&D ευθύνη. Μ' αρέσουν λέξεις όπω η ευθύνη. Ε, εμείς ε, προβληματιζόμαστε. Η πρόταση του κυρίου, των κυρίων Φερχόστατ και Μπρόκ πιστεύουμε ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση και μας αρέσει που ε, πολλές προτάσεις επιτροπής του κύριου Κάσμαρακ παραδείγματος χάρη έχουν ληφθεί υπόψη αλλά εκρεμεί ένα σημαντικότατο ζήτημα ποιος έχει την τελική ευθύνη την τελική ηγετική θέση για την ανάπτυξη η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν από ποιον θα ηγείται για τα αναπτυξιακά ζητήματα. Κάπου μέσα στο κείμενό σας κύριοι θα ήθελα να αναφέρετε αυτό. Ε, το ίδιο και στην πρόταση της κυρίας Άστον. Δηλαδή μια ειλικρινή έκκληση ε, ε, για το άρθρο 208 της Συνθήκης Λισαβόνας όπου προβλέπεται ότι πρέπει να υπάρχει ό,τι γίνεται στα πλαίσια της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης πρέπει να είναι συνεκτικό σε σχέση με τους αναπτυξιακούς μας στόχους. Ποιοι είναι αυτοί, βιώσιμη ε, μείωση μάλλον της ε, φτώχειας με βιώσιμο τρόπο. Ε, ό,τι δεν ευθυγραμμίζεται με την βιώσιμη εκρίζωση της στόχιας τελικά δεν συνάδει με τη συνθήκη. Μπορούμε να τα πούμε έτσι, να τα πούμε αλλιώς, να εφεύρουμε συνέχεια νέες δομές αν θέλετε, αλλά πρέπει να οργανωθούμε από κοινού γιατί αλλιώς σημαίνει ότι δεν παίρνουμε ούτε τη συνθήκη στα σοβαρά. Εγώ θέλω να μιλήσω για την πολιτική βούληση ελπίζω να ε, τύχω υποστήριξη. Πολιτική βούληση λοιπόν, ούτω ώστε ε, να προωθηθούν τα αναπτυξιακά ζητήματα ε, χωρίς να το ρηψοκινδυνεύσουμε ότι οι ιδέες μας για την ε, αναπτυξιακή βοήθεια θα ε, χρησιμοποιηθούν για σκοπιμό της εξωτερικής πολιτικής. Δεν ταυτίζονται τα δύο απαραίτητα. εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμη πώς ο κύριος Πίμπαλξ θα μεριμνήσει ώστε όσοι δραστηριοποιούνται επιτόπου τόπου στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κάνουν αυτό που προτείνεται ε, στην αναπτυξιακή πολιτική αν πρέπει να περάσουν όλα αυτά από την κυρία Άστον. Ε, θα πάνε από τη γάμα δέλτα από τον Πίμπαλξε, μετά θα περάσει το θέμα από την Άστον και μετά θα επιστρέψει στις επιτόπου αντιπροσωπείες. Ε, υπάρχει εγκάρση ευθύνη δηλαδή εν τη αυτή περιπτώση και θα ήθελε η Επιτροπή και το Συμβουλίο να μου απαντήσουν και οι κύριοι Μπρό και Φερχόφστατ που δεν ε, ενέκριναν μία πρόταση του κυρίου Κάσμαρακα, δηλαδή για τη συνολική διευθέτηση διαφορών μέσα στο Συμβούλιο, με εξηγήσουν γιατί δεν το έκαναν. Ευχαριστώ. Κύριος Γκερέρο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν είναι αλήθεια ότι η σοκολάτα βοηθάει για να μας φτιάχνει τη διάθεση σαφέστατα, αυτό που είναι γεγονός θα έπρεπε να είχαμε έρθει με γενναία δόση και απόθεμα σοκολάτας. Έχω ακούσει επανειλημμένα και τον κύριο Μπροκ και τον κύριο Φερχόφστατ, γιατί είμαι και μέλος της Επιτροπής ε, ε, ε, Συνταγματικών Υποθέσεων. Και έχω την εντύπωση, θα ήθελα να με διαψεύσουν, θα το επιθυμούσα, αλλά έχω την εντύπωση ότι σήμερα είναι η μέρα που τους είδα πιο απεσιόδοξους από όλες ή να απέχουν περισσότερο από την συνάντηση με την πρόταση της ΥΠΑΤΗΣ ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ο κύριος Φερχόφστα διακόπτηκε. και εκτός μικροφώνου παντά κιόλας. Λοιπόν, δεν πέφτω και πολύ έξω από ό,τι φαίνεται λοιπόν σε αυτά που λέω. Νομίζω ότι ε, υπάρχει εξή διπλός κίνδυνος και απορρέουν αυτά από τα όσα ακούσαμε και από τον κύριο Φερχόφστατ κύριος. Ο πρώτος κίνδυνος είναι η εξωτερική πολιτική της Ένωσης την οποία ουσιαστικά υπομίζεται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να περιοριστεί αν δεν συμφωνήσουμε και να αναχθεί μόνο στην ασφάλεια, την άμυνα, τη διπλωματική δράση και να απαγκιστρωθεί τελείως η ανάπτυξη, η γειτονία, η ανθρωπιστική δράση. Νομίζω ότι αυτό είναι κίνδυνος και θα πρέπει εν πάση ε, περιπτώσει και πάση θυσία να αποφευθεί. Δεύτερος κίνδυνος. Ως Συνέπεια αυτού, η αναπτυξιακή πολιτική να μην καταλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συνεπώς να επιστρέψουμε σε κατάσταση τύπου της σημερινής. Μα δεν γίνεται αυτό. Γιατί αλλάζουν όλα τα υπόλοιπα. Είναι αδύνατο να παραμείνουμε στη σημερινή κατάσταση για την αναπτυξιακή πολιτική. Τη στιγμή που το θεσμικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος της Ένωσης και η φιλοδοξία της στην εξωτερική πολιτική διαφέρουν. Έχουν αλλάξει. Τώρα, πώς θα αποφύγουμε αυτούς τους δύο κινδύνους. Νομίζω ότι η εστίαση που μας παρουσιάσατε είναι η σωστή. Δεν μπαίνω σε πιο ειδικά θέματα, γιατί δεν είμαι κυμπεριγνώμων βέβαια. Αλλά πώς θα αποφύγουμε αυτό το δεύτερο κίνδυνο. Και τους δύο κινδύνους μάλλον. Η εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα η λειτουργία της Επιτροπής αυτής, της δράσης, θα πρέπει να είναι μια υπηρεσία που να έχει στρατηγική, μεγάλες κατευθύνσεις γραμμές και στόχους συγκεκριμένους και να ενώνει. Και αυτά όλα να ε, καθορίζονται από τους επιτρόπους μαζί με την ύπατη εκπρόσωπο υπό τη σαφή της ηγεσία αλλά με ε, άμεση συμμετοχή ε, των Επιτρόπων Ανάπτυξης, Γειτονίας, Ανθρωπιστικής Δράσης κτλ. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος εξωτερικής πολιτικής τη Ένωση, ποιε είναι οι μεγάλες κατευθυντήριε γραμμές, οι στρατηγικέ δράσει, τελικοί, οι βασικοί στόχοι, να συμμετέχουν στην κατάρτιση όλων αυτών και στην χάραξη της πολιτικής και οι αρμόδιοι επίτροποι για τα επιμέρους χαρτοφυλάκια. Και ως συνέπεια όλων αυτών εκ των υστέρων το επίπεδο ευθύνης και αυτονομίας στην εκτέλεση των πολιτικών ανάπτυξης ανθρωπιστικής δράσης και γειτονίας να αναλογεί κυρίως στους επιτρόπους και στις δομές που σήμερα εξαρτώνται από αυτούς. Δηλαδή, θα πρέπει να αποφύγουμε αυτή την αποσύνδεση που μας είπε ο Φερχόφστατ. Για την πρώτη επιλογή που νομίζω ότι σωστά την κατάλαβα. Στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον καθορισμό των στόχων να συμμετέχουν οι επιτροποί και άρα να θεωρείται κοινοτική πολιτική αυτή με κοινοτικό προϋπολογισμό σαφέστατα Αυτό θα πρέπει να γίνει για να αποφύγουμε τη δεύτερη επιλογή που θα ήταν όλεθρο και για την εξωτερική πολιτική και για την αναπτυξιακή πολιτική. Γιατί ούτε η εξωτερική πολιτική θα ήταν ισχυρή και συνεκτική χωρίς την ανάπτυξη, ούτε η, Επιτροπή ανάπτυξη, η ε, πολιτική ανάπτυξη τη της Ευρωπαϊκής αν αποσυνδεθεί από την εξωτερική πολιτική. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτά που άκουσα από τους πρώτους ομιλητές δεν με καθησυχάζουν. Οι διαφορές ε, εντός των θεσμικών οργάνων ε, παραμένουν. Το ειδικό καθεστώς της υπηρεσίας αυτής είναι αμφίσιμο, γι' αυτό πρέπει να υπαγρυπνούμε κάτι διάρκεια εφαρμογής ε, και δημιουργίας της νέας υπηρεσίας. Το πρόγραμμα της κυρίας Άστον που παρουσιάστηκε δημιούργησε διαφορετικές αντιδράσεις στο Συμβούλιο ε, σε σχέση με την πολιτική ανάπτυξη σε αυτή τη νέα θεσμική δομή. Γι' αυτό πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η εξωτερική υπηρεσία δεν είναι πολιτικό όργανο λήψη αποφάσεων, αλλά είναι μια υπηρεσία που βοηθάει την ύπατη εκπρόσωπο ε, για την άσκηση των καθηκόντων της ε, στα πλαίσια της εντολής της. Ε, λόγω του οργανογράμματος και των ε, εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και των θέσεων που δημιουργούνται, πιστεύουμε θα δημιουργούν ε, πάρα πολλές συγκρούσεις που θα υπέσκαπταν το στόχο αυτής της υπηρεσίας. Πώς να μην είμαστε ανήσυχοι με την ιδέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ο ένας από τους βοηθούς της ΥΠΑ της εκπροσώπου είναι ανατίθεται στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Οι σοσιαλιστές δεν είναι υπέρ του διορισμού ενός βοηθού της ύπαρξης εκπροσώπου ε, που να βασίζεται στο μέλημα για πολιτική ισορροπία. Σε ό,τι αφορά την οργάνωση της υπηρεσίας, η κυρία Άστον έκανε τη συμβολική επιλογή να εγκαταστήσει το γραφείο της στο εσωτερικό της Κομισιόν, αλλά έχει ένα τριπλό, μια τριπλή ιδιότητα που είναι ιδιάζουσα είναι αντιπρόεδρος τη Κομισιόν και άρα έχει αρμοδιότητα για τι αρμόδιε αρχέ για τι εξωτερικέ υποθέσει, αλλά δεν υπόκειται στη συλλογικότητα ε, της Κομισιόν ε, ή στην εξουσία του Προέδρου της Κομισιόν. Τι σχέσει θα έχει η στην εξουσια του προεδρου τη κομισιον τι σχεσει θα εχει η κομισιον και η Εξωτερική Υπηρεσία, η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ποιε γενικέ ε, ε, διευθύνσει θα ενταχθούν στη νέα υπηρεσία. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξη τι ρόλο θα έχει και πώ ο ρόλο τη ανάπτυξη ε, θα ληφθεί επαρκώ υπόψη στα διάφορα επίπεδα προγραμματισμού της ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση των τομεακών πολιτικών σε αυτή τη νέα υπηρεσία, το θέμα της ενσωμάτωση της πολιτικής ανάπτυξης σε αυτή τη νέα υπηρεσία είναι κρίσιμης σημασίας. Η ομάδα μας ε, θέλει η υπεύθυνοι και οι ευθύνε των κάθε επιτρόπων να μην επηρεαστούν από τη δημιουργία αυτή τη υπηρεσία εξωτερική δράση. Οι πολιτικέ αποφάσει θα πρέπει να εξακολουθούν να λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω καθορίζεται στην συνθήκη τη Λισαβόνα. Εξάλλου, είναι σημαντικό να υπάρχει μια συνέπεια και συνεκτικότητα ανάμεσα στον προγραμματισμό τη εξωτερική βοήθεια και τη εφαρμογή τη. Γι' αυτό τα προνόμια της θα πρέπει να εξακολουθούν να εξαρτώνται από την ευθύνη των αρμοδίων ε, επιτρόπων για να υπάρχει μια συνέχεια ανάμεσα στους πολιτικούς στόχους και στην εφαρμογή τους επιτόπου. Επίσης, ε, το σχέδιο της κυρίας Άστον δεν είναι αρκετά σαφές και ενεργές σε ό,τι αφορά την ε, διπλή κλίδα. Και στο Λουξεμβούργο δεν έχει χυθεί άπλετο φως από το θέμα θα πρέπει η προσέγγιση να διευκρινιστεί, ούτω ώστε στην περίπτωση της κοινή μεικτής αρμοδιότητας, ο αρμόδιος επίτροπος να διατυπώνει πολιτικές που θα παρουσιάζονται από κοινού από τον Επίτροπο και τον Αντιπρόεδρο ή ύπατη εκπρόσωπο στο Σώμα των Επιτρόπων. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε για το ρόλο του Επιτρόπου ε, ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να υποστηρίξουμε την συμπερίληψη της ανθρωπιστικής βοήθειας στο, στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης, ενώ αυτό το θέμα δεν είναι πολιτικό. Ε, είναι ένα ερώτημα θεμητό να τεθεί. Η εξωτερική δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πρέπει να έχει έτσι και συνέπεια και ορατότητα. Η συνέπεια είναι πολύ σημαντική. Είναι σημαντικό για να υπάρχει εμπιστοσύνη από τους εταίρους μας ε, και εμπιστοσύνη και από τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Η κυρία Τσίμερ. Α, τώρα λειτουργεί. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι συνάδελφοι μου μίλησαν εκτενώς για τα θέματα που μας απασχολούσαν τους τελευταίους μήνες και εβδομάδες ε, σε σχέση με την ε, ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Θα ήθελα να προσθέσω δύο λεπτομέρειες για να μην επιμηκύνω. Το πρώτο επιχείρημα για ποιο λόγο έχουμε τέτοιες επιφυλάξεις ότι η αναπτυξιακή πολιτική τελικά δεν λειτουργεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει υπό την ηγεσία ενός διπλωματικού σώματος. Στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουμε δει και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέχρι σήμερα. Χωρίς ε, εντολή ε, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν μπορούν να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι για την καταπολέμηση της στόχιας και οι καθυστερήσει στην ανάπτυξη. Αν δεν υπάρχει σαφής αναπτυξιακή εντολή. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εδώ ε, βρίσκεται σε ένα τεράστιο δίλημα λειτουργικό και θα πρέπει να λυθεί. Για να λυθεί αυτό θα πρέπει να έχει επιτέλους ε, αντίστοιχη εντολή από αρμόδιο πρόσωπο και υπό την αιγίδα της εξωτερικής ε, πολιτικής δεν μπορεί αυτό να λειτουργήσει. Και ένα δεύτερο που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Οι μελέτες που υπάρχουν, οι γνωμοδοτήσεις ξέρω εγώ, αναφέρουν αυτά τα στοιχεία. Η πρώτη της κυρίας Άστον ε, φέρεται να έρχεται σε αντίφαση με το άρθρο 208 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την αναπτυξιακή βοήθεια. Στόχος μας είναι η μείωση της στόχης και η τελική εκρίζωση της στόχιας. Αυτό ε, είναι δεσμευτικό, είναι πρωτογενές δίκαιο η συνθήκη δηλαδή για όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν μπορεί κανείς αυτό να το αντιπαρέρχεται χωρίς τροποποίηση της συνθήκης επειδή έτσι θέλει να κατατάξει κάπου την αναπτυξιακή πολιτική. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αν έχει ληφθεί αυτό επαρκώς υπόψη ή αν δεν έπαιξε κανένα ρόλο στη συζήτηση. Ευχαριστούμε ο κύριος Ευχαριστώ πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ τους κυρίους Μπρό και Φερχόφστατ. Πάω στην καρδιά του θέματος. Ε, έπρεπε να πάω στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Μπορεί να επαναλάβω κάποια πράγματα. Εφόσον δεν έχουμε χρόνο, με διακόψετε άμα τα έχουν πει άλλοι. Λοιπόν, λέει εδώ financial tools, χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Ε, τι πιστεύετε κύριε για την τροπολογία μας. Λέμε εδώ ότι ο προγραμματισμός ε, θα πρέπει να συμφωνηθεί από κοινού από τον αρμόδιο επίτροπο και την ύπατη εκπρόσωπο. Είναι λογική η πρότασή μας και σε τι χρησιμεύει, εν πάση περιπτώσει, η υπηρεσία εξωτερική δράση για να έχουμε αυξημένη διαφάνεια και για να έχουμε καλύτερε συνέργειε, καλύτερη συνεργασία. Αλλά ε, η τροπολογία μας δεν αντιβαίνει στο διτό αυτό στόχο. Εμείς επιθυμούμε μέσα από την τροπολογία να έχουμε μεγαλύτερη συνοχή. Αλλά αυτό δεν ε, αντιβαίνει το, σε αυτό το διπλό στόχο που έλεγα. Μεγαλύτερη διαφάνεια δηλαδή και καλύτερη συνεργασία. Ε, ούτως ή στην πράξη έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Αν θέλουμε καλύτερη συνεργασία, ας έχουμε ε, τα απαιτούμενα μέσα στη διάθεσή μας. Ε, ας φροντίσουμε να τα έχουμε. Δηλαδή θα έχουμε πράγματα στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης που δεν θα είναι υπό την αρμοδιότητα του κυρίου Πίμπαλξ. Κακοφωνία θα έχουμε. Δεν θα έχουμε καλύτερη συνεργασία αν συμβαίνει αυτό. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Ε, θα ήθελα να προσπογράψετε αυτή τη θέση γιατί κατά αυτόν τον τρόπο ε, θα ενισχύσετε και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιον του Συμβουλίου, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε η κυρία Κέλλερ τώρα. Το μεσημέρι κάναμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση όχι στην Επιτροπή, έτσι, σε ένα άλλο κύκλο για την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης με τον κύριο Κριστόφερσον, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Είναι ένας από τους ε, λίγους συμβούλους της κυρίας Άστον ε, για την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Εγώ τρόμαξα με τη συζήτηση, να σας πω την αλήθεια. Ούτε καν σκέφτηκαν τους ε, μηχανισμούς για την ανάπτυξη αυτής της πολιτικής και ούτε συζητούν για το πώς θα βελτιώσουν τη συνεργασία και τον συντονισμό των δωρητών, ούτε για το πώς ε, θα έχουν τον κύριο λόγο οι δικαιούχες χώρες, πώς θα βελτιωθεί όλη αυτή η προσπάθεια. Όχι απάντηση δόθηκε, ούτε σκέψη δεν έχει αφιερώσει σε αυτό. Και είπε ότι ο μόνος μηχανισμός που υπάρχει είναι το άρθρο 208 και ωραίο που το έχουμε, αλλά κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει και κάτι άλλο για να προσφέρει κανείς στο δικαστήριο όταν βλέπει ε, κάποιες ε, ασυνέπειες στην πολιτική. Και κάτι άλλο που δεν είναι σαφές είναι ότι κάποιες αρμοδιότητες αναπτυξιακής πολιτικής στην ομάδα της κυρίας Άστον ε, θα ε, ορίζουν ποια θα είναι η δική μας αναπτυξιακή πολιτική. Καλό είναι να έχει κανείς ιδέες και πολύ χρήσιμο να ακούς και απόψεις έξωθεν, αλλά Μήπως να ακούσουν και κανέναν που έχει και αρμοδιότητα και δουλεύει και χρόνια στο χώρο, να ακούει και εμπειρίες ε, που έχουν αποκομίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένη δεκαετίες ολόκληρες στην αναπτυξιακή συνεργασία. Χρειαζόμαστε και ένα ισχυρό λόμπι για τα συμφέροντα της ανάπτυξης, γιατί δεν ταυτίζονται πάντα με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτά ε, δεν τα έχουν χωνέψει αυτοί που έχουν την αρμοδιότητα να τα ασκούν ως πολιτικοί. Και για την πρότασή σας, είπαν και συνάδελφοι, τελικά παραμένει το ερώτημα για τη διαπραγμάτευση με την κυρία Άστον. Το δικό της έγγραφο θα διαπραγματευτούμε, όχι το δικό σας. Ποια από τα θέματα αυτά λοιπόν είναι δική σας προτεραιότητα και το απορρίπτει η κυρία Άστον και θα συνεχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε γι' αυτό, να το καταγγέλουμε ή θα επικεντρωθούμε κάπου αλλού και ποια θα είναι η θέση μας. Έχουμε και ανταλλάγματα εκεί για τη διαπραγμάτευση, για παζάρι. Ευχαριστώ αγαπητοί κύριοι βουλευτές. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εν συνεχεία πίσω πάλι στον κύριο Μπροκ και στον κύριο Φερχόστατ για να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ε, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη, πολύ σύντομα, γιατί δεν θέλω να ξοδέψουμε πολύ χρόνο στην απάντηση. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο κύριος Γκερέρο σε μεγάλο βαθμό. Ε, η αμοιβαία α, βοήθεια μεταξύ εξωτερικής πολιτικής και αναπτυξιακής πολιτικής δημιουργεί μια δυναμική ε, αυτό θα προωθήσει τις πολιτικές και θα βασιζόμαστε λιγότερο στα διάφορα μέσα και εργαλεία. Ο κύριος Τιγολιά είπε το εξής. Ε, η συζήτηση ε, μερικές φορές έχει πάρει λάθρος ε, δρόμο. Ε, αν είναι πολιτικό σώμα αυτό ή θεσμικό σώμα. Είναι μια υπηρεσία, ούτε το ένα είναι, ούτε το άλλο και δουλεύει υπό την πολιτική ευθύνη της ε, Επιτροπής Ανάπτυξης. Εκτός μικροφώνου τα σχόλια. Για την ανάπτυξη, άρθρο 8, που λέει ξεκάθαρα ότι υπό την άμεση εποπτεία και καθοδήγηση με αυτόν τον τρόπο κάθε υπηρεσία κάθε τεχνική υπηρεσία δουλεύει για έναν επίτροπο. Και εγώ. Ε, και στρεφόμαστε προς τους επιτρόπους ε, για πολιτική καθοδήγηση. Στο άρθρο 8 ε, μιλάμε για θεματικό προγραμματισμό. Αλλά δεν μιλάμε καν για άμεση μιλάμε για υποπτία. Ας μην παίζουμε με τις λέξεις. Η πολιτική ευθύνη για την έναξη ε, του προγραμματισμού, για την δημιουργία των στρατηγικών εγγράφων ε, αναχώρα για την εφαρμογή υπάρχει. Και ο Επίτροπος Ανάπτυξης, ο προγραμματισμός, όλες οι χώρες, για τον προγραμματισμό των χωρών και την εφαρμογή ε, των προγραμμάτων για όλες τις χώρες. Ε, επομένως, ε, οι αρμοδιότητες είναι ξεκάθαρες. Υπάρχει και ρόλος και ευθύνη του Επιτρόπου Πίμπαλξ στην χρήση των πόρων EAS τεχνικών πόρων για να κάνει την ε, δουλειά του, την πολιτική δουλειά ε, για την οποία είναι υπεύθυνη ενώπιόν σα. Και αυτό το λέει το κείμενο. Τρίτον, το Συμβούλιο στην Πολιτική Συμφωνία ε, απέρριψε την ιδέα ενός πολιτικού βοηθού ή ιονή πολιτικού βοηθού της, είπα, της εκπροσώπου για την νομιμότητα όλων των θεμάτων Συμφωνώ με αυτά που είπε για την περιγραφή του άρθρου 21. Αν είναι κάτι παράνομο, ε, θα πρέπει να το καταδείξουμε. Τέταρτον, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές που αποφασίζονται από τον κύριο Πίμπαλξ εφαρμόζονται συνεχεία. Ένα άλλο άρθρο λέει ότι η επικεφαλής αντιπροσωπείας λαμβάνει οδηγίες από όλους τους αρμόδιους επιτρόπους. Πολιτική καθοδήγηση. Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του Επιτρόπου Πίμπαλξ και του ε, επικεφαλής αντιπροσωπείας που βρίσκεται στη χώρα. Ε, και από την ύπατη εκπρόσωπο λοιπόν και από κάθε επίτροπο που έχει ευθύνη. Το λέει αυτό το άρθρο. Τέλος. Το θέμα της πολιτικής συνέπειας και της εξάλληψης της φτώχειας. Θα εκφραστεί μέσω της πρότασης για τα, που κάνουμε για τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα και τα στρατηγικά έγγραφα αναχώρα, ε, τα οποία υπόκεινται και τα δύο στον έλεγχό σας. Είναι... μπορείτε να τα σταματήσετε. Αυτά θα τα προτείνει ο Πίμπαλξ και επομένως έχετε τη ε, δυνατότητα να ασκήσετε το δημοκρατικό σας έλεγχο. Ελπίζω στο μέλλον όλη αυτή η πρόταση να βοηθήσει για να μεταφράσουμε όλα αυτά σε υποχρεώσεις στον προϋπολογισμό. Και τώρα ε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπρόκ για να απαντήσει τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να μια παρατήρηση. Η υπηρεσία αυτή ε, είναι ε, έχει ως στόχο μάλλον να ε, συνενώσει δύο πράγματα που είχαν διαφορετικές νομικές βάσεις. Η ΚΕΠΑ που τελικά πάει στο Συμβούλιο και τα υπόλοιπα εξωτερικά θέματα. Αυτά τα λέγει το άρθρο 17 της Συνθήκης. Εκτός της ΚΕΠΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει την εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαφές είναι αυτό στην Επιτροπή είναι η αρμοδιότητα για όλους τους τομείς τελικά και θα πρέπει να προσέξουμε ε, στην αρχιτεκτονική αυτής της υπηρεσίας, στην κατασκευή και όπως είπε σωστά ε, κάποιος συνάδελφος είναι υπηρεσία και δεν είναι όργανο λήψης αποφάσεων να μην έχει de facto ε, μεγαλύτερο βάρος η διακυβερνητική συνεργασία και να είναι μόνο στα χαρτιά η δυνατότητα λήψης αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλωστε, γι' αυτό θέλουμε κι εμείς να τονίσουμε τους ε, επιτρόπους στην πρότασή μας και να τους φέρουμε στο προσκήνιο. Η πολιτική εκπροσώπηση αλλά και η διαβούλευση είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εκεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πώς έχουν τα πράγματα. Σε περίπτωση σύγκρουσης, αυτός που θα πρέπει να πάρει την απόφαση είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Άστον ηγείται της ΚΕΠΑ, αλλά στα υπόλοιπα θέματα συνεισφέρει στην ΚΕΠΑ ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν προσπαθούν να βρουν λοιπόν κάποια συνοχή, αλλά υπάρξει μια σύγκρουση μεταξύ του Αρμοδίου Επιτρόπου και της κυρίας Άστον, αποφασίζει το σύνολο, το σώμα των Επιτρόπων και ουδής άλλος. Δεν έχει η ίδια αρμοδιότητα λήψη αποφάσεων η κυρία Άστον πάνω από τον άλλο επίτροπο που διαφωνεί μαζί τη. Και αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να ισχύσει και στην πράξη. Καταλαβαίνω ότι δεν αρέσουν οι της ε, στον κύριο Κάσμαν. γιατί πριν από λίγο καιρό ανήθηκε να είναι Πάπας και ο ίδιος, γιατί και ο Πάπα κάποιο πρόσωπο είναι πηγή. Κάτι λέει ο κύριος Κάσμαν, δυστυχώ δεν τον ακούμε. Ε, έλεγα λοιπόν, δεν του αρέσουν οι αναπληρωτές του κυρίου Κάσμα, ντέπιουτης αυτή. Ε, αλλά το, το είπε και ο κύριος Μπέρμαν, σε περίπτωση σύγκρουσης αποφασίζει το σύνολο των επιτρόπων, το σώμα των επιτρόπων που είναι αρμόδιο κατά τη συνθήκη. Για ΚΕΠΑ, και μόνο για την ΚΕΠΑ είναι αρμόδιο το Συμβούλιο, για όλα τα υπόλοιπα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι λύνονται και πολλά ερωτήματα και απορίες για το ποιος έχει την ηγεσία. Και ε, ε, το ρώτησαν και πολλοί συνάδελφοι. Και επειδή ο ύπατος εκπρόσωπος είναι και αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής δεν μπορεί να τα κάνει μόνα του όλα αυτά και να προτείνει σε συνεργασία με τον Επίτροπο Ανάπτυξη. Σήμερα δεν μπορεί να αποφασίσει κανένα επίτροπο τίποτα από μόνο του για δεσμευτικέ αποφάσει νομοθετικέ και τέτοια. Είναι συλλογικό σώμα η Επιτροπή. Οπότε σε αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Θα πρέπει να φροντίσει να βρει βέβαια και την πλειοψηφία για τι θέσει του. Όπω κάνει και σήμερα ο κάθε επίτροπο. Έτσι δεν είναι. Και θα πρέπει να το προσέξουμε και αυτό. Άλλο θέμα πώς έχει η αλυσίδα της διοίκησης, η δομή της διοίκησης, chain of command. Με τον ίδιο τρόπο και στις εθνικές κυβερνήσεις το ίδιο είναι. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται ο καθένας αρμόδιος να δίνει μια οδηγία εντολή ή διαταγή στον κάθε πρέσβη σε περίπτωση μια μιας θεομηνίας. Χαθήκαμε αν γίνει αυτό θα πρέπει πάντα να πηγαίνει μέσω ε, της κυρίας Άστον και των επικεφαλής αντιπροσωπείας και τα λοιπά. Αλλά ε, ε, γνώση των αρμοδίων να γίνεται αυτό. Παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα που δεν το γράφει πουθενά. Εμπόριο. Αν ο αρμόδιος για το εμπόριο επίτροπος δώσει μια εντολή και το μπλοκάρει, είπατε, εκπρόσωπος ή αντιπροσωπεία, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να αποφασίσει το σώμα των επιτρόπων για τις εντολές και τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελεστούν. Σήμερα αυτό είναι στα χέρια των εθνικών κυβερνήσεων. Ας πούμε, ο οικονομικός εμπορικός ακόλουθος είναι από το Υπουργείο Εμπορίου. και αν έχουν διένεξη ο Υπουργό Οικονομικών με το Υπουργό Εξωτερικών και δεν διαβραστεί αυτή η εντολή στην πρεσβεία, αποφασίζει η κυβέρνηση. Αλλά δεν θα πηγαίνει ο καθένα, ξέρω εγώ, Υπουργό να διατάζει τον τάδε ακόλουθο και τον δίνα. Αυτό θα γίνει γελιογραφία, καρικατούρα για τον υπόλοιπο κόσμο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και θα αρχίσει ο κάθε υψηλό βαθμός υπάλληλο να δίνει εντολές και οδηγίες στη διπλωματική υπηρεσία και θα έχουμε το απόλυτο χάος και για όλα τα θέματα. Λοιπόν, πιστεύω ότι αν γίνει αυτό έτσι κύριε Γκερέρο, δεν θα είμαι τόσο απεσιόδοξος για την πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Ούτε πρόκειται να κυριαρχήσει και να καταπιεί όλα τα άλλα και να τα... καθό αντίστροφο θα έβλεπα εγώ. Διότι σε σχέση με την υπηρεσία αυτή εξωτερικής δράσης, ορισμένα θέματα της ΚΕΠΑ δεν είναι άμεσα ε, ε, υπαγόμενα στο Συμβούλιο, αλλά ε, παρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Attached to the Commission το λένε αυτό. Και αυτό είναι ενδιαφέρον και από τη σκοπιά του Κοινοβουλίου. Να ασχοληθείτε και από αυτή τη σκοπιά Δηλαδή, αν φανούμε εξύπνοι εδώ, μπορούμε να το αντιστρέψουμε και να το εκμεταλλευτούμε γι' αυτό. Ας έχουμε λοιπόν λίγο περισσότερο θάρρος. Αν θέλουμε ε, αυτό να γίνει συνεκτική πολιτική και συνεπής, για τη διαχείριση των κρίσεων, ως παράδειγμα, Γιατί ε, ε, θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις σε συμβούλια που να συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι μόνο στρατιωτικοί και αυτό ε, τονίζει περισσότερο την πρόληψη από ότι τη στρατιωτική επέμβαση, όπως προβλέπει άλλωστε και η συνθήκη. Και μια τέτοια εξέλιξη νομίζω θα μπορούσαμε να την αξιοποιήσουμε, να την εκμεταλλευτούμε για να προχωρήσουμε. Και στο προγραμματισμό, κύριε Γκέρενς. Και η κυρία Τσίμερ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και βέβαια αυτό πάντα είναι ένα θέμα τι πολιτικές επιθυμίες έχει ο καθένας. Ένα πλαίσιο και μόνο είναι και η συνθήκη της Λισαβόνας. Ένα μέσο είναι ε, ε, αυτή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Τώρα, το πώς χρησιμοποιείς αυτό το μέσο και το εργαλείο εξαρτάται από τις πολιτικές πλειοψηφίες και τους πολιτικούς συσχετισμούς κάθε φορά και το κέντρο βάρους και τις προτεραιότητες. Και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό ούτε στο μέλλον. Δεν μπορούμε να ορίσουμε συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους από το γεγονός ότι ιδρύουμε μια νέα υπηρεσία ή έχουμε μια πρωτογενή συνθήκη. Σε τελική ανάλυση εκλογές αποφασίζουν το σχετισμό της πλειοψηφίας. Σύντομος θα είμαι, Πρόεδρε. Ο κ. Μπρόκ εξήγησε πολύ καλά τη λογική της πρότασής μας. Και τελικά, στη λογική της πρότασής μας, όλα απόκεινται στην απόφαση του Σώματος των Επιτρόπων. Αν υπάρχει διαφορά, διένεξη για την εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής. Εξακολουθώ να πιστεύω φυσικά ότι η πρόταση της κυρίας Άστον έχει τον κίνδυνο ότι δημιουργεί μια έλλειψη συνέπειας και συνεκτικότητας γιατί χωρίζει τα γεωγραφικά από τα θεματικά θέματα. Μπορούμε να πούμε ότι η ιεραρχία είναι η ίδια, αλλά είναι δύο διαφορετικές προτάσεις. Την πρόταση Άστον, όπου η υπηρεσία εξωτερικής δράσης δεν συνδέεται με την Κομισιόν, δεν εντάσσεται στην Κομισιόν και αποτελεί ένα φορέα εντελώς ανεξάρτητο. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στον προπολογισμό Όλες οι δράσεις κανονικά της ε, Ένωσης είναι στο κεφάλαιο 3, στο κοινοτικό κεφάλαιο, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως, η μάχη που δίνουμε εγώ και ο Μπροκ είναι να αλλάξει αυτό και να πούμε ότι αν θέλουμε να δώσουμε ειδικέ εγγυήσεις γιατί το Συμβούλιο ε, θέλει να κάνει εξωτερική πολιτική, με ειδικέ εγγύησει. Γι' αυτό θα πρέπει τα, γεωγραφικά desk τα οποία θα διαχειριστούν την ανάπτυξη θα φτάσουν σε ένα άλλο κεφάλαιο του προϋπολογισμού διαφορετικό από τις Κομισιόν. Και η Κομισιόν θα κάνει τον προγραμματισμό σε θεματικό και οριζόντιο επίπεδο. Ε, γίνεται αυτή η διάκριση. Πρέπει να συνεχιστεί η μάχη λοιπόν για το θέμα αυτό. Άκουσα πολλούς που γνωρίζουν από αυτά τα πράγματα ε, και άκουσα και από μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκφράζουν αμφιβολίες για το τελικό αποτέλεσμα που πετύχαμε από τους επιτρόπους για την πρόταση αυτή. Ορισμένοι λένε, ας έχει το Κοινοβούλιο, ας αμφισβητήσει την απόφαση που ελήφθη. Στρεφόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή τώρα για να προασπιστεί τις, ε, τα προνόμια και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Α, δεν συμβαίνει για πρώτη φορά, ε, μην νομίζετε. Δεύτερον, το άρθρο 208 αυτό υπάρχει στο κείμενο, το δικό μας κείμενο. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι το συντομότερο δυνατό να δείτε και εσείς τις τροπολογίες που η Επιτροπή ΑΦΚΟ και η Επιτροπή ΑΦΕΤ ε, παρουσιάζουν. Που θέλουν να εσωματωθεί το άρθρο 208 της συνθήκης, να ληφθεί υπόψη και τι σχέση πρέπει να υπάρχει μεταξύ της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αναπτυξιακής πολιτικής και της πολιτικής συνεργασίας. Ορισμένε ιδέες δεν υπάρχουν. Παραδείγματο χάρη στο κείμενό μας λέμε ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, και οι αρμόδιες επιτροπές της ε, οι αρμόδιες συγγνώμη, υπηρεσίες της Επιτροπής θέλετε να βάλετε εσείς. Για μας δεν υπάρχει διαφορά γιατί για μας στην εξωτερική υπηρεσία ε, είναι και οι υπηρεσίες προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΒΕ υπό την αιγίδα του Επιτρόπου. Του Επιτρόπου και ο Επίτροπος Ανάπτυξης είναι αναπόσπαστο τμήμα της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης μαζί με την ύπατη εκπρόσωπο. Και όταν υπάρχει πρόβλημα διαφοράς και σύγκρουση μεταξύ των δύο, το σώμα των Επιτρόπων αποφασίζει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάσμα θέλει να εκφράσει, να μιλήσει για αυτό τα συμπεράσματά του. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω θερμά αυτούς που πήραν το λόγο και συμμετείχαν στη συζήτηση. Μια συζήτηση σημαντική. Οι δύο παρεμβάσεις των δύο συνεισηγητών ε, θεωρώ ότι ήταν πολύ αισιόδοξε. Γιατί μιλάνε για μια συνένεση για τις, ε, και λένε ότι οι υπηρεσίε ε, εξωτερικής δράση δεν θα είναι ούτε ένα θεσμικό όργανο, ούτε ένα ιονή θεσμικό όργανο, γιατί δεν υπάρχει βάση στη συνθήκη. Και αφού δεν θα είναι θεσμικό όργανο, αποκλείεται να μειωθεί ο ρόλος των επιτρόπων και η σημασία της αναπτυξιακής πολιτικής. Αυτό που φοβόμαστε περισσότερο για τη σημασία της πολιτικής ανάπτυξης είναι ο, είναι ο ρόλος της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Ελπίζω να διατηρηθεί και ελπίζω να καταλήξουμε σε συνένεση. Ευχαριστώ λοιπόν τους δύο εισηγητές. για να είμαστε σαφείς, για να ε, μην υπάρχει καμία παρανόηση. Ο Γκί και ο Έλμαρ να, ε, ε, να υπολογίσω ότι θα υιοθετήσουν την τροπολογία μας για τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Από ό,τι κατάλαβα συμφωνείτε απολύτως μαζί μας. Παραφράσατε τη θέση μας όταν πήρατε το λόγο πριν ε, λήξει συνεδρίας να υποθέσω ότι ε, υπάρχει ομοθυμία. Ναι ή όχι. Μικρόφωνο γιατί δεν ακούμε τι λέει ο κύριος Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο δικό μας κείμενο και το δικό σας. Διαβάσαμε τα δύο κείμενα εδώ. Τι προσθέτετε εσείς. Ε, κάθε φορά που λέμε εμείς η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, εσείς προσθέτετε και την Αράδα και οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μα εννοείται ότι για μα εννοείται, εξπακούεται ότι ε, ε, εντάσσονται οι υπόλοιπε υπηρεσίες στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Έχουμε διαφορετικό εφαλτήριο σε σχέση με την Άστον. Ε, ας το δούμε διμερώς, αν χρειάζεται τροποποίηση, αν ναι, κανένα πρόβλημα. Η Europaid θα κάνει την υλοποίηση και στις δύο περιπτώσεις, έτσι, για την αναπτυξιακή πολιτική θα εκτελέσει την αναπτυξιακή πολιτική. Και δεν υπάρχει ε, καμία αμφιβολία σχετικά με το ότι το σώμα των Επιτρόπων θα αποφασίσει. Η Επιτροπή έχει τον τελευταίο λόγο. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία λοιπόν. Ναι, δεν υπάρχει, Σάγλε, καμία παρανόηση. Μην ανησυχείς. Ευχαριστούμε τους συναδέλφου. Ε, ευχαριστούμε κύριε Φερχόφστατ, κύριε Μπρόκ. Έχουμε άλλο ένα σημείο. Κύριε Μπέργκμαν.